We finished earlier after the trade partnership and uh, Giacolino. Ladies, gentlemen, colleagues. Uh, Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να αρχίσουμε, είναι 9 και 10 και είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα. Let's uh, start our meeting. Αρχίζει λοιπόν η συνεδρίαση. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Προτείνω δύο αλλαγέ. Το 18 και το 24 αναβάλλονται για μια επόμενη συνεδρίαση. Το 18 αφορά την έκθεση για την Κίνα και ζητάω η, η εισηγήτρια μάλλον η κυρία Ντοσαρνέζ να αναβληθεί η συζήτηση και η ψηφοφορία, καθώς και το 24, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Ο κύριος Καμάλης, ηγητής λοιπόν, ζήτησε να αναβληθεί επίσης η συζήτηση. Τώρα, παρά το γεγονός ότι αφαιρούμε αυτά τα δύο θέματα από την ημερήσια διάταξη, έχουμε παρόλα αυτά 24 σημεία τα οποία πρέπει να συζητήσουμε συμπεριλαμβανομένης και της ανταλλαγής απόψεων με τον ε, Πασκαλαμή. Ε, επίσης έχουμε ακρόαση με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Ντεκούχτο, την συνεδρίαση των συντονιστών. Άρα θα πρέπει να τηρούμε το χρόνο που έχει προβλεφθεί για τη συζήτηση κάθε θέματος πρακτικά τις συνεδρίες του Ιανουαρίου τα έχετε λάβει. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις ή σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Όπως ξέρετε, μεταδίδεται απευθείας από το ίντερνετ η συνεδρίαση, εξαιρουμένη της συνάντηση των συντονιστών. Σας έχουν ε, διανεμηθεί οι επιστολές που έχουν ανταλλαγεί. Αν κάποιος ε, ζητά κάτι άλλο, η γραμματεία στη διάθεση. Τώρα, περνούμε. Στο επόμενο θέμα. Έχουμε ένα νέο μέλος στην Επιτροπή μας, την κυρία Μπαντία. Σας καλωσορίζουμε. Έρχεσαι από μία από τις ε, πιο πολύ άσχολες επιτροπές, σε μία από τις πιο πολύ άσχολες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, το πρώτο σημαντικό μας θέμα, η πρόοδος των τριμερών διαπραγματεύσεων. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία συζητώνται αυτή τη στιγμή αφορά τον κανονισμό για τις ε, συμβάσεις ξένων επενδύσεων. Εγώ είμαι συγγετής Χθες Είχαμε την πέμπτη συνάντηση τριμερών διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και έχω καλά νέα να σας πω. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με όλα αυτά τα θέματα, έγινε διάλογος λοιπόν με την Δανική Προεδρία για πρώτη φορά έδειξε μια κάποια ευελιξία το Συμβούλιο και τη βούληση να προχωρήσει και να καταλήξει σε συμβαστικές λύσεις με το Κοινοβούλιο. Υποβάλαμε μια προσφορά εμείς εκ μέρους μας και η ανταπόκριση του Συμβουλίου για πρώτη φορά δεν ήταν αρνητική. Συμφωνήσαμε λοιπόν να ζητήσουμε την Επιτροπή να έρθει σε επαφή με το Συμβούλιο για να προσπαθήσει να βρει μια κάποια ισορροπία μεταξύ των θέσεων των δύο μερών και να καταλήξει σε μια συμβαστική πρόταση αποδεκτή από όλους. Δεν έχουμε ακόμη για την επόμενη συνάντηση ημερομηνία. Θέλω να ελπίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε όταν θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο θέμα αυτό, διότι έχουμε καθυστερήσει. Monitoring ε, activities of monitoring groups. Since our last meeting, a number of um, το επόμενο θέμα είναι το 5, δραστηριότητα της εποπτικής ομάδας. Ο Τζον Λούκας είναι ο εισηγητής για το θέμα του Μερκοσούρ, δεν είναι παρόν. Ο Παύλο Θάλβα είναι επίσης συγγετής για την Κεντρική Αμερική. Η κυρία Κορέια όμως θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος του κύριου Παύλου Ασάλδα, ο οποίος μου ζήτησε σήμερα πολύ σύντομα να σας εξηγήσω τι έγινε χθε στη συνάντηση της Εποπτικής Ομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Αμερικής. Εχθές στις 28 Φεβρουαρίου συναντήθηκε για δεύτερη φορά η εποπτική ομάδα για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και είχαμε και την παρουσία των πρέσβων της Γουατεμάλας, ο εκπρόσωπος σε θέματα εμπορίου ήταν παρόν, Νικαράγουα, Ψεβεδατόρ, Ονδούρα, Κωνσταντίνα και Παναμά. Μαζί με τον κύριο Σάλβα, τον κύριο Λάγκεν που εκπροσωπούσε τον κύριο Λέμφλι, τον σκιαδησηγητή και τον κύριο Σόφτ, καθώς και εκπρόσωποι των διάφορων πολιτικών ομάδων ήταν παρόντος. Ο κύριος Θάλμπα ευθύς εξ αρχής είπε πόσο σημαντικά από εμπορικής πολιτικής και συνεργασίας θα είναι αυτή η πρώτη συμφωνία περιφερειακής, περιφερειακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κεντρική Αμερική. Παρουσίασε την εμπορική πτυχή για θέματα ανάπτυξης και ενσωμάτωσης που προβλέπονται και για τα δύο μέρη στη συμφωνία. Τις ίδιες απόψεις εκφράσαν και οι πρέσβεις, μεταξύ των οποίων ο πρέσβης Κωνσταντίνο και είπε ότι η συμφωνία αυτή είναι πραγματικά ένας στόχος με τον οποίο θα υπάρξει σταθερότητα και βελτίωση των σχέσεων και των δύο μετών. Και τα δύο συμβαλόμενα μέρη είπαν πόσο τους ενδιαφέρει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε και είπαν ότι θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Καταρχάς προβλέπεται να αποφασίσει το Συμβούλιο για την υπογραφή του το Μάιο, ώστε μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να το εγκρίνει. Από τη μεριά τους οι πρέσβεις ε, δεν ανέφεραν ότι υπάρχει πρόβλημα με την επικύρωση σε εσωτερικό επίπεδο και τους ενδιαφέρει η δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής του τετάρτου μέρους που αφορά τα εμπορικά θέματα. Θα πρόκειται για μικρή ε, συμφωνία με ε, κοινά υποχρεώσεις για όλους τους αλλά χρειάζεται και από εμάς η επικύρωση. Κυρίως όσον αφορά το σημείο 4, υπάρχουν πλεονεκτήματα για τις άμεσες επενδύσεις και για να ανοίξουν οι αγορές για μας. Τελικά είπαμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία υπογραφή αυτή της συμφωνίας και τα δύο μέρη, κυρίως σε εμπορικό επίπεδο, δεδομένου ότι θα είναι μια υποδειγματική διμερής συμφωνία ε, για πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι τώρα για την ε, εργασία που επιτελεί, η εποπτική ομάδα. Υπάρχουν κάποιες εξελίσεις. Εγώ είμαι εισηγητής για την θέματα με τη ΣΥΠΑ. Είχα με την ε, ε, αμερικανική πλευρά σε θέματα εξωτερικού εμπορίου μία συνάντηση και τα άλλα τα μέρη της ομάδας της υποπτικής γνωρίζουν ποιες ήταν οι απόψεις που εκφράστηκαν από τον ε, εκπρόσωπο των ε, Αμερικανών ε, επιχειρηματιών στην Ευρώπη. Εκουαδόρ και Βολιβία. Επίσης έγινε συνάντηση συγητής όμως Σόλτς, ο οποίος δεν είναι παρόν. Είπαν ότι ο Μαρτίν Καζάκα θα ήθελε επίσης να πει κάτι για την δική του την ομάδα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Είχαμε την πρώτη συνάντηση υποπτικής μας ομάδας Ευρωπαϊκής Ένωση Ιαπωνίας αυτό το μήνα και, οργανώσαμε, και συζητήσαμε θέματα οργανωτικά. Συναντιόμαστε τέσσερις φορές το χρόνο και με την παρουσία διαφόρων ενδιαφερομένων ε, μέρους της Ιαπωνίας και δική από την Επιτροπή έκανε μία σύντομη παρουσίαση της προόδου που επιτελείται και θα κάνει ένα ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Στο ψήφισμα αυτό θα υπάρξει η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ε, αρχή διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι όλες οι συζητήσεις αυτές θα τελειώσουν το τέλος Μαρτίου, δεδομένου ότι μας πιέζει η Ιαπωνία, δεδομένου ότι υπάρχουν ε, κρεμοί ακόμη τα θέματα της Κορέας και της ε, καταστροφής της Περσινής. Ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις που εκφράστηκαν από την αρχή. Συζητήκαμε τον Οκτώβριο του 2011 για θέματα ε, κρατικών προμηθειών και άλλα θέματα. Πιστεύουμε ότι στον τομέα αυτό έχουν βρεθεί επιτυχείς λύσεις και οι διαπραγματεύσεις για τα θέματα αυτά των πολυμερών διαπραγματεύσεων και θέματα κρατικών προμηθειών έχουν προχωρήσει. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε με τις συναντήσεις της υποπτικής ομάδας και θα παρακολουθούμε την πρόοδο η οποία υπάρχει στις ε, συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Έχετε την εντύπωση ότι θα είναι ε, ε, θετικές οι εξελίξεις. Ναι, ναι, ναι. Ζητήσαμε και από την Επιτροπή να μας πει ποια είναι η δική της αξιολόγηση και νομίζω ότι μπορώ να πω ότι είναι μετρίως αισιόδεξη. Πολύ διπλωματικά αυτά τα οποία λέτε για το θέμα αυτό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στο σημείο 6 τώρα. Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλία. Ο εισηγητής είναι ο Μυροσλάβ Ράντσντορφ. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με τους περισσότερους εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης τέτοιου είδους συμφωνίες με στόχο να ε, κάνουμε κάποιες ε, ε, συμβάσεις που θα αφορούν περιοχές ελεύθερου εμπορίου με τις με περισσότερες χώρες. Έχετε το λόγο κύριε Ράντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αλλά αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των εμπορικών μας σχέσεων με την ε, ε, ανατολική πλευρά της Υπήρου αυτής. Θεωρώ ότι ορισμένοι δεν γνωρίζουν ότι οι ανατολικές συνεργασίες περιλαμβάνουν ε, έξι χώρες οι οποίες ανήκουν στην ανατολική στην ανατολική πλευρά και ε, περιλαμβάνουν το Αζερβαϊτζάν, την Αρμανία, την Μολδαβία, την Γεωργία και την Ουκρανία. Ε, υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση εκτός από την Λευκορωσία και αυτές οι συμφωνίες σύνδεσεως περιλαμβάνουν μια πολύ σημαντική συμφωνία η οποία αποβλέπει σε, στη δημιουργία ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών όχι μόνο από πλευράς δασμολογικής αλλά και από πλευράς του κοινοτικού κεκτημένου και ε, αποβλέπουν και στην κατάργηση των ε, μη δασμολογικών εμποδίων για τη διεξαγωγή του εμπορίου. Ε, όσον αφορά τώρα την Ουκρανία. οι συμφωνίες και συζητήσεις για την ε, DC38 ε, έχουν ολοκληρωθεί ε, ορισμένες άλλες συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Ουκρανία και πιστεύω ότι οι συμφωνίες δεν θα πρέπει να είναι όμοιροι αυτών των περιορισμών και γι' αυτό προτείνω να υπάρξει μία προσωρινή εφαρμογή της DCFTA για να προωθήσουμε το εμπόριο και ε, έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα στην Ουκρανία και να προωθεί τις αναγκαίες ε, πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες ε, που μπορούν να βοηθηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι στο τελευταίο ταξίδι στην Ουκρανία επισκέφθηκα τεράστιες επιχειρήσεις, μία που παράγει ε, ε, ε, βλήματα που έχει 2.000 εργαζομένους είναι ένα πολύ σύγχρονο εργοστάσιο το οποίο όμως δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία παραγγελία και μπορεί να βοηθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη γεωργία και την ε, Μολδαβία που περιλαμβάνονται στις ε, συζητήσεις αυτές και τις διαπραγματεύσεις CFTA οι οποίες ε, έχουν ξεκινήσει και πρέπει να διεξαχθούν τις επόμενες ε, εβδομάδες για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν χωρίς ε, καθυστερήσεις. Το πρόβλημα της ε, Μολδαβίας είναι πολιτικό. και αναφέρεται ε, εις ε, ε, την κατάσταση του, της εδαφικής κυριαρχίας διότι υπάρχει ένας υψηλός αριθμός στρατιωτικών που δεν έχουν όμως τόσο σημαντικό ρόλο στη χώρα όσο στο παρελθόν. Τα προβλήματα όμως παραμένουν και η κεντρική κυβέρνηση της ε, γεωργίας ε, ε, ελέγχει μόνο τον πυρήνα της χώρας παρόλο που έχουν γίνει οικονομικοί πρόοδοι ιδίως στον ενεργειακό τομέα και εφόσον ε, έλαβαν πιστώσεις μπόρεσαν ε, να ξεκινήσουν ε, μικρά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγά και να εξάγουν ηλεκτρισμό στα γειτονικά κράτη δηλαδή βλέπουμε κάποιες πρόοδους. Όσον αφορά την Αρμενία, ε, ξεκινήσαμε τις ε, συζητήσεις CFTA μόνο αφού μεταφράστηκε η έκθεση μου και ε, γι' αυτό το τμήμα που αναφέρεται σε αυτή τη χώρα της έκθεσής μου πρέπει να προσαρμοστεί και να αντικατοπτρίζει την ε, πρόσφατη κατάσταση και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα με βοηθήσουν με ορισμένες τροπολογίες ε, να προβώ σε αυτή την ενημέρωση. Προσβλέπω λοιπόν στη συζήτηση και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να με βοηθήσετε για να βελτιώσω την έκθεσή μου. Θέλω επίσης να σας πω ότι στην ε, πρώτη ανταλλαγή. Η Επιτροπή μας είπε ότι η αρχή των διαπραγματεύσεων του CFTA με την ε, Αρμενία δεν ε, θα ξεκινούσε ε, σύντομα. Δύο μήνες όμως μετά ξεκίνησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις χωρίς να δοθεί καμία ένδειξη στην Επιτροπή Ίντα. Ελπίζω λοιπόν ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αλληλέγγυα μαζί μας. και ότι θα να μας ενημερώνουν γέρος και πλήρως θα προβαίνουν σε μια ελημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμερίζονται ε, τις πληροφορίες που έχουν κατά τρόπον ώστε και εμείς να μπορούμε να περιλαμβάνουμε τις σημαντικές εξελίξεις και να τις σημειώνουμε και να τις περιλαμβάνουμε στις περαιτέρω δραστηριότητές μας όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν το Αζερβαϊτζάν σήμερα αντιπροσωπεύει 70% ε, του ΑΕΠ των χωρών του Καυκάσου. Δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη οικονομική επίδοση των χωρών αυτών έχει μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη λόγω <clears throat> του πετρελαϊκού τομέα και μετά από την ιστορική συμφωνία μεταξύ του κράτους του Αζερβαϊτζάν και των μεγάλων εταιριών πετρελαίου μπόρεσαν να προχωρήσουν και στην έκθεση μου ενθαρρύνω το Αζερβαϊτζάν να να διαφοροποιήσει την οικονομία της χώρας και να προσβλέπει σε μία συμμετοχή εις τον ΠΟΕ για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Αζερβαϊτζάν και ε, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη περίπτωση στην έκθεση αυτή είναι η Λευκορωσία. Διότι όπως γνωρίζετε υπάρχουν ορισμένα πολιτικά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Λευκορωσίας καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατακρίνει σταθερά την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Λευκορωσίας και πιστεύω ότι αυτή η σχετική απομόνωση της χώρας δεν είναι παραγωγική για το μέλλον διότι άλλοι οικονομικοί παίκτες είναι έτοιμοι να εισέλθουν στην Λευκορωσία όπως οι Κινέζοι παραδείγματος χάρη και με την στάση της η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπορεί να υποφεληθεί ε, από τις δυνατότητες αυτής της χώρας και δεδομένης ε, της κατάστασης της Λευκορωσίας εάν την εξετάσουμε αντικειμενικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένας σταθερός οικονομικός και πολιτικός ε, συνεργάτης, ότι η κατάσταση είναι καλύτερη από την Ουκρανία, ότι οι επιχειρήσεις υπάρχουν, παράγουν και εξάγουν και ε, το ηθικό της Λευκορωσίας είναι υψηλό και γι' αυτό θεωρείται ένας σταθερός συνεργάτης. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα που υπάρχουν με τη Λευκορωσία και να μην συνεχίσουμε με αυτή τη στάση η οποία απομονώνει την ε, χώρα αυτή. διότι μέσω της οικονομικής συνεργασίας μπορούμε να προωθήσουμε την ε, κατάσταση, μπορούμε να προωθήσουμε ε, και ε, την κατάσταση της μεσαίας τάξεως της Λευκορωσίας κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να προωθηθεί η κοινωνία των πολιτών και ε, να προκαλέσουμε μεγαλύτερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις τις οποίες προσβλέπουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την άνοιξη του 2011 αυτή η ε, ανατολική τέρη ίσως ε, κάπως παρέμεινε στο περιθώριο λόγω των εξελίξεων στο νότιο χώρο και τώρα τα μέσα ενημέρωσης στρέφουν το βλέμμα τους και πάλι από τους νότιους εταίρους και στρέφονται προς ανατολικά. Πιστεύω λοιπόν ότι η ευημερία των ανατολικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι σημαντική ε, για την ενότητα της Υπήρου μας και ε, ήταν αντιπαραγωγικό το ότι παραμελήσαμε αυτούς τους εταίρους μας στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις ε, εμπορικές σχέσεις με αυτούς και επίσης είναι σημαντικό να προωθήσουμε τις πολιτικές ε, ε, δραστηριότητες ε, μαζί τους. Έχω ε, εστιαστεί στα εμπορικά θέματα στην έκθεσή μου και πιστεύω ότι υπάρχει μία καλή βάση για συζήτηση και προσβλέπω στα σχόλιά σας ε, και νέες ιδέες που μπορούν να συμπεριληφθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Ράνστορφ. Ε, η έκθεσή σας είναι πιο εκτενής από ό,τι συνήθως αλλά αντιλαμβάνομαι την σημασία και το θέμα αυτό ο όντως είναι σημαντικό. Πρέπει επίσης να σας πω ότι έχω λάβει μία επιστολή από ένα μέλος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που ξέχασα αυτή την πληροφορία και δεν την ανέφερα γιατί όντως έχουμε λάβει τα σχόλια του κυρίου Όλεκ Λιάσκου, μέλους ε, του Ουκρανικού Κοινοβουλίου ο οποίος μας είπε ότι τον ικανοποιεί η έκθεσή μου. Ας προχωρήσουμε τώρα εις ε, τους σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Κούτας εφόσον δεν είναι ο κύριος Ζελέσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο που εκπώνησε. Η έκθεση είναι μακροσκελής, αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά ολοκληρωμένη και εξισορροπημένη. Όπως είπε ο εισηγητής, ε, τα γεγονότα και εξελίξεις ε, στη Βόρεια Αφρική έχουν ε, μεταφέρει το επίκεντρο της προσοχής μας Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσέχουμε περισσότερο τους ε, νότιους γείτονές μας, αλλά θα πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τους ανατολικούς εταίρους μας. Δεν θέλουμε να αμελήσουμε αυτή την πτυχή της ε, πολιτικής γειτονίας μας. Άλλος μεγάλος στόχος πρέπει να είναι η καταπολέμηση και εξάλληψη της ε, φτώχειας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε την σταθερότητα στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Γιατί ο δημοκρατισμός αυτών των χωρών εξαρτάται άμεσα και συνδέεται άμεσα με ε, το, την αύξηση του βιωτικού επίπεδου, τη διασφάλιση της ελευθεροτυπίας, ε, την ενδυνάμωση των ε, ίδιων των δημοκρατικών θεσμών. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές πτυχές της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συμφωνώ πολύ με τον εισηγητή η κοινωνία των πολιτών μπορεί πράγματι να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο ε, σε ό,τι αφορά τα μακροπρόθεσμα ωφέλη. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούμε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ευρωπαϊκή αγορά για τους ε, ανατολικούς εταίρους. Αφού αναφερθήκατε στη Μολδαβία, 47% των εξαγωγών της Μολδαβίας ε, κατευθύνονται προς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντική η επιρροή μας, λοιπόν. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω εδώ και θα το συμπεριλάβω και σε τροπολογίε είναι η ανάγκη εισαγωγή ενό κεφαλαίου για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. στι συμβάσει ελεύθερων συναλλαγών, ελεύθερων εμπορίου ε, με τι χώρε τη Ανατολική Εταιρική Σχέση. Αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον εισηγητή και ε, στο τέλο θα έχουμε μια εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ. Άλλοι όχι. Ας περάσουμε σε μέλη της Επιτροπής. Η Θέλερ. Ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένιωθα λίγο αόρατος Η μια στιγμή. Νομίζω ο Πρόεδρος, εγώ μίλησα για τους ε, σκιώδεις. Νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία του κ. Ράνστοφ. Ιδίω το σχέδιο έκθεσης για τις χώρες και αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ σημαντική αυτή η προσθήκη. Αναγνωρίζεται την κατάσταση στην Λευκορωσία. Αποτελεί ενδεχομένω τη μεγαλύτερη πρόκληση ανάμεσα σε αυτές τις χώρες της περιφέρειας. Παρόλο που η έκθεση ε, στηρίζει απολύτως τις διμερείς ε, διαπραγματεύσεις σε πέντε από τις έξι χώρες, για μας δεν καθορίζει πραγματικά τον στόχο ε, αυτής της σύμβασης ελεύθερων συναλλαγών. Μιλά για οικονομική ενσωμάτωση και ρυθμιστική σύγκληση, αλλά δεν παρέχει κάποιο μέτρο σύγκρισης ε, για, να μπορέσουμε να, να μετρήσουμε, αν θέλετε, την, ε, την πρόοδο που σημειώνεται για να αποφασίσουμε αν όσα έχουν γίνει είναι αρκετά. Μία από τις πηγές έμπνευσης αυτής της έκθεσης ήταν η κοινή ανακοίνωση Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, της είπα εκπροσώπου εξωτερικών σχέσεων. Και εκεί υπαριθμόν ένα στόχος αυτής της συμφωνίας ήταν η, πραγματική δημοκρατία. Μια δημοκρατία που λειτουργεί ε, με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με κράτος δικαίου. Όλα αυτά είναι θεμελιώδεις πυλώνες ε, της εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ε, εταίρους Αυτή είναι η πρώτη μας φιλοδοξία. Η δεύτερη φιλοδοξία είναι η καθιέρωση στενότερων ε, δεσμών με την κοινωνία των πολιτών, που θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τον πρώτο στόχο, να επιτύχουμε τον πρώτο στόχο. Αλλά εγώ δεν βλέπω αρκετή τεκμηρίωση, αν θέλετε, στην έκθεσή σας για αυτές τι πτυχέ. Δεν μας παρέχει δηλαδή αυτή η έκθεση τα εργαλεία και τα μέσα που χρειαζόμαστε για να αξιολογήσουμε την ε, πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ε, πολλοί από αυτού τους ανατολικούς εταίρους διαθέτουν οικονομικές δομέ που θα πρέπει να ανεκοδομηθούν για να ε, αντικατοπτρίζουμε καλύτερο τρόπο τις προτεραιότητες της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι η ενσωμάτωση αυτών των χωρών είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση για να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή σε αυτές τις χώρες. Και εγώ λοιπόν θέλω να ε, συμβάλλω περαιτέρω στην ανάπτυξη και διαμορφούση αυτή τη έκθεση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ακούγοντα τα όσα είπατε, είδα ότι τίτλος της έκθεσης είναι οι εμπορικές πτυχέ τη ανατολική εταιρική σχέσης, όχι οι πτυχέ τη εξωτερική πολιτική. Τώρα, ας ακούσουμε την κυρία Τζικόφσκα από την Επιτροπή. Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή επικροτεί αυτή την έκθεση για τις εμπορικές στοιχείες της Ανατολικής Τερικής Σχέσης. Είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένη ε, αυτή η έκθεση και ε, εντοπίζει τις μεγαλύτερες ε, προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας ό,τι αφορά την Ανατολική Εταιρική Σχέση στον τομέα του εμπορίου. Το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο τη Ανατολική τερική Σχέση, καθώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων τη Ανατολική τερική Σχέση, την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ενσωμάτωση η ολοκλήρωση. Μέσω αυτών των εμπορικών συμβάσεων θα ε, παράσχουμε στους ανατολικούς εταίρους μας πλήρη ε, πρόσβαση στην ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς, χωρίς τρευλώσεις για να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους ε, και την ανάπτυξή τους. Ως αντάλλαγμα ζητούμε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για αυτές τις χώρες προκειμένου να υποφεληθούν ε, ε, πλήρως των ευεργετημάτων που τους προσφέρουμε. Η Επιτροπή στηρίζει απολύτως αυτή την ε, ατζέντα και την ε, προωθούμε. Το 2011 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και η συμφωνία με την... έχει συναυθεί η συμφωνία με την ε, Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να οριστικοποιήσουμε το κείμενο. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ της Συμφωνίας Σύνδεσης και της CFTA είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτό θα πρέπει να ε, ε, πληρώνονται σημαντικοί όροι για να επωφελούνται αυτά τα κάτι μελη της ε, εμπορικής συμφωνίας. Θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μια ενιαία θέση σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία και τη Μολδαβία, αυτές οι χώρες έχουν σημειώσει σημαντική και ουσιαστική πρόοδο στις προσπάθειές τους ε, να εφαρμόσουν ε, θεμελιώδεις ε, μεταρρυθμίσεις. Έχει δοθεί το πράσινο φως από τα κρατημέλη βάσει έκθεσης της Επιτροπής, την οποία μοιραστήκαμε μαζί σας, όπου δεσμευθήκαμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία. Και το 2012 Έχουμε προγραμματίσει ε, εντατικές διαπραγματεύσεις σε τέσσερις γύρους και ο Επίτροπος του Γιούχτ αυτή τη στιγμή επισκέπτεται αυτές τις δύο χώρες για να ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο τις διαπραγματεύσεις. Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων θα λάβει χώρα, χώρα στις 3, θα τέλει Μαρτίου, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά την Αρμενία. Έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τη Γεωργία και τη Μολδαβία. εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε στενά μαζί με αυτή τη χώρα. Στα τέλη του 2011 η κυβέρνηση οθέτησε ένα πολύ φιλόδοξο ε, σχέδιο δράσης για να είναι έτοιμοι μέχρι τα τέλη του 2011 και κατάφεραν να πετύχουν ε, τους στόχους ε, που είχαν θέσει. Στις 17 Φεβρουαρίου τα κράτη-μέλη και πάλι βάσει έκθεσης της Επιτροπής ε, που μοιραστήκαμε μαζί σας αποφάσισε να στηρίξει την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την ε, Αρμενία. Ε, αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το τεχνικό προπαρασκευαστικό έργο για να προετοιμαστεί το πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσει φέτος το σημαντικό δυνατόν. Για τις υπόλοιπες χώρες, είναι απαραίτητη η ε, συμμόρφωση με τις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, των μελών του ΠΟΕ για αυτές τις χώρες, κυρίως το Αζερβαϊτζάν και τη Λευκορωσία. Το Αζερβαϊτζάν δεν είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΠΟΕ, αλλά θα συνεχίσουμε να προωθούμε την ενδυνάμωση των σχέσεων με αυτή τη χώρα στο πλαίσιο και των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία, για τη Λευκορωσία ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή πρέπει να γίνει μέλος του ΠΟΕ. Μια μελλοντική προτιμησιακή συμφωνία θα πρέπει να αποτελεί τμήμα μια ε, συμφωνία σύνδεση. Και όπω ξέρετε, μια συμφωνία σύνδεση μπορεί να συναυθεί βάσει ε, κοινών ε, αξιών. Δυστυχώ δεν συμμεριζόμαστε τι ίδιε αξίε με τη Λευκορωσία όμω. Θα τελειώσω σε δύο λεπτά. Αυτό που είναι σημαντικό με αυτέ τι χώρε είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και η Επιτροπή σας θα είναι πλήρως ενήμερη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Επαναρχόμαστε στον εισηγητή για μια σύντομη σύνοψη, γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα πριν περάσουμε στον Πασκάλεμι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου και την εκπρόσωπο της Επιτροπής για τις παρατηρήσεις τους για το θέμα της κοινωνίας των πολιτών. Και ο κύριος Κιούτας και ο κύριος Τέιλερ αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι το στοιχείο κλειδί της ε, στρατηγικής να ενδυναμώσουμε την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να υπάρξει σύγκληση μεταξύ Ανατολικής Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι κάποιες μέθοδοι είναι εύκολο να προωθηθούν για να ενδυναμώσουν την κοινωνία των πολιτών. Για παράδειγμα, να τους βοηθήσουμε στην, στην βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησής τους. Τα δικά μας ευρωπαϊκά πρότυπα μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε αυτές τις κοινωνίες. Σε ορισμένες ε, γειτονικές χώρες υπάρχουν προγράμματα για την προώθηση τέτοια της διαδικασίας, αλλά θα πρέπει να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες και να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διοικητικές δομές λοιπόν πολύ εύκολα μπορούν να βελτιωθούν, δεν είναι τόσο δαπανηρό. Επίσης, ε, σε κάποιες στοιχείες της λειτουργίας της, του επιχειρηματικού κόσμου θα πρέπει να εισαγαγούμε πιο ανεπτυγμένες μορφές λογιστικής, για παράδειγμα, που είναι ιδιαίτερα παροχημένες ορισμένες από τις ε, ανατολικές χώρες. Ένα-δυο στοιχεία ανέφερα μόνο, αλλά Νομίζω ότι το κύριο μέσο είναι η ενδυνάμωση, για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών είναι οι εμπορικές σχέσεις. Όταν συζητήσαμε το θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, αυτό είναι κάτι που παίρνει χρόνο. Νομίζω ότι στην αλληλουχία των σταδίων πρώτα απ' όλα έρχεται το κράτος δικαίου. Γιατί αυτό οδηγεί στην εγκαθίδρυση της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι, προέρχεται από την, από την πρακτική μας εμπειρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ελπίζω να με βοηθήσετε να τροποποιήσω την έκθεση μέσω τροπολογιών. Γιατί στην περίπτωση της Αρμενίας υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις μετά την ε, μετάφραση. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες μέχρι την 21η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Περνούμε στο σημείο 7. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. Ε, ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας από την ΕΝΒΗ. Έχουμε γνωμοδότηση από τον συγκητή Σαλβατόρα Γιακολίνο. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος διότι Ήδη έχουμε εξετάσει αυτόν τον φάκελο και ουσιαστικά πρέπει να διατυπώσουμε μία γνωμοδότηση για ένα θέμα πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρεται στην αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ε, υπάρχουν ε, νέες δυνατότητες για να υπάρχει μία βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της πράσινης τεχνολογίας για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αλλά και με εμπορικές συμφωνίες οι οποίες να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Στα πλαίσια της, των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ε, έχουμε και καλές περιβαλλοντολογικές σχέσεις γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ενταθεί η διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό και υπενθυμίζω εδώ το, τη συμφωνία της ΔΟΑ ε, για τις δασμολογικές και μη δασμολογικές προόδους ε, που έχουν μεγάλη σημασία σε αυτό το πλαίσιο πλαίσιο. Όσον αφορά, όσον αφορά την, ε, ε, την ε, ε, ε, ε, βιωσιμότητα πρέπει να ανοίξουμε και μία νέα πτυχή δηλαδή να μπορέσουμε να καλύψουμε τους, τα μέσα παραγωγής να συνδυάσουμε τα περιβαλλοντολογικά με τα εμπορικά μέτρα και να συντονίσουμε τις διάφορες ενέργειες οι οποίες πρέπει να συνάδουν με τις σημαντικές αλλαγές που διαπιστώνουμε στην κοινωνία. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξουν δασμολογικές προτιμήσεις για τα οικολογικά προϊόντα ε, στο σύστημα. Αυτό θα αποτελούσε μία προστιθέμενη αξία στις ε, σχέσεις με τις υποανάπτυξη χώρες ιδίως εάν σκεφτούμε το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Ευρώπη για το 2020. Πρόκειται εδώ για ένα θέμα το οποίο είναι στη διάθεσή σας, ένα κείμενο το οποίο μπορεί να βελτιωθεί και αυτά θα πω μόνο τώρα και στη συνέχεια κατόπιν από τα σχόλια των συναδέλφων της Επιτροπής μπορώ να επανέλθω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε με τους σκιώδης, ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο για μια πολύ καλή πρόταση. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την περιβαλλοντική πτυχή, γιατί όλα αυτά ε, συμβάλλουν και στην αηφόρα ανάπτυξη. Ε, το δίκαιο και βιώσιμο εμπόριο θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των εμπορικών μας πολιτικών. Γι' αυτό και χαιρετίζω την ε, πρότασή σας να και να προσθέσουμε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρόταση στις υφιστάμενες συμφωνίες θα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο οικουμενικό σύστημα για την δίκαιη αξιοποίηση των ε, πόρων μας, πάντα σε συμμόρφωση και με, τον, με τα πρότυπα του ΠΟΕ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έλλειψη συνοχής σε ό,τι αφορά τη δέσμευση της δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί ενώπιον του ΠΟΕ και του, του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Γι' αυτό θέλω να συμβάλλω στην ε, γνωμοδότησή σας με τις ε, δικές μου ιδέες και προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία μαζί σας. Κάθριν Ευχαριστώ, Κάθριν Μπίρντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομη. Θέλω να χαιρετήσω κι εγώ αυτή την γνωμοδότηση. Είναι καλή, καλύπτει πολλά στοιχεία. Στην πρώτη παράγραφο λέτε ότι μπορεί να είναι, να είναι αηφόρος, πρέπει να το τονίσουμε λίγο. Has to be, θα πρέπει να είναι αηφόρος, γιατί αν δεν είναι τότε δεν υπάρχει εμπόριο. Ίσως θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι εδώ για την ασφάλεια τροφίμων. Γιατί η εμπορία φυσικών πόρων είναι σημαντική. Χθε ο ΠΟΕ ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο για την επιστηστική ασφάλεια στο μέλλον. Και αυτό, καθώς θα, θα περνάει ο καιρός, θα γίνει το λένε και πιο σημαντικό. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος, ότι θα πρέπει το εμπόριό μας να είναι δίκαιο και αηφόρο και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ε, που έχουν διαμορφώσει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το εμπόριο δεν θα πρέπει να ε, εμποδίζει τις χώρες αυτές ε, να αναπτύσσουν τους τη δική τους εμπορική δραστηριότητα. Επίσης, οι πράσινες τεχνολογίες. Βλέπουμε μη δεσμολογικά εμπόδια να ανακύπτουν. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τα όσα κάνουμε σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Γιατί πρέπει να προσέχουμε αυτό το ζήτημα με θεωρήσεις και άλλα εμπόδια ε, που ανακύπτουν. Και αυτό το say what you pay, κάτι που έχουν υιοθετήσει τώρα οι Αμερικανοί, θα πρέπει και εμείς να το ενσωματώσουμε στις μελλοντικές μας εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Um, Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος δηλαδή να ε, ακολουθήσω το σχόλιο της Κάθριν ο οποίος είπε ότι το δίκαιο εμπόλιο πρέπει να είναι βιώσιμο διότι διαφορετικά δεν είναι δίκαιο. Γι' αυτό και έτσι χαιρετίζω την έκθεση και τον εισηγητή ο οποίος ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση βεβαίως όμως τα προβλήματα ε, συνήθως ε, ε, βρίσκονται στις λεπτομέρειες. Όταν δηλαδή μιλάμε για περιβαλλοντολογικά προϊόντα και αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να δούμε και την οντότητα των επιχειρήσεων που παράγουν αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Δηλαδή η ηλιακή ενέργεια στη Γερμανία είναι πολύ ε, προχωρημένη στο διεθνή ανταγωνισμό. Πρέπει να δούμε δηλαδή με ποιον τρόπο θα προωθήσουμε τα διάφορα αυτά αγαθά. Και εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ε, ε, το, στην παράγραφο 3 την, ε, για το Ρίο 20 την οποία προετοιμάζομαι για την, ε, τον επόμενο γύρο που θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δούμε τι έχει ήδη συμφωνηθεί στο θέμα αυτό. Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες ε, θα έπρεπε να προσθέσουμε ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύουν τις περιβαλλοντολογικές ε, απόψεις για όλα τα θέματα και να θυμηθούμε ότι τα περιβαλλοντολογικά και τα οικονομικά θέματα είναι συνδεδεμένα διότι αν ε, δεν κινούμεθα σε μία κοινωνική πραγματικότητα τότε ε, έχουμε ξεπεράσει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και κάποια ε, ευθύνη θα πρέπει να αναφέρεται στο σημείο αυτό, ότι έχουμε δηλαδή κάποια ευθύνη. Και ε, προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία με τον εισηγητή στο θέμα αυτό. Τέλος ο Κίθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαι εγώ σκιώδης, αλλά μου έχει αφήσει τις ε, σημειώσεις του ο συνάδελφος. Θέλετε να συνεχίσω. Σχέδιο γνωμοδότησης εστιάζεται κυρίως στην ε, άνοιγμα των ε, διεθνών αγορών για θέματα εμπορίου και υπηρεσιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για ανοιχτέ αγορέ για τι εξαγωγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλε χώρε. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται ότι λείπει είναι το άλλο μίση του εμπορίου. Η διάσταση των εισαγωγών που είναι η Ήπειρος, η Ευρώπη όπως ξέρουμε είναι η Ήπειρος που εξαρτάται στα μεταργίες περισσότερο από Και από τα περισσότερα τα οποία πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μία ε, φυή και σε θέματα ενέργειας κοινωνική πολιτική. Όλοι υποστηρίζουν την αηφορία, πράγμα που σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει πραγματικά να αποσυνδέσουμε την οικονομική ανάπτυξη από την αυξημένη χρησιμοποίηση πόρων. Και αυτό είναι κάτω με την εξοικονόμηση ενέργεια, την χρησιμοποίηση ενεργειακών προϊόντων ανακύρωση και την χρησιμοποίηση αρχών για την εξοικονόμηση ενέργειας. Νομίζω ότι μπορούμε να προσβλέψουμε σε συνεργασία με τον εισηγητή για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάποιες νέες ιδέες, να καταθέσουμε τροπολογίες σε θέματα σχέσεων, σε θέματα ε, νέων κανονισμών για τα ενεργειακά. Και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται για η αηφόρο εμπόριο. Θα θέλαμε επίσης η Επιτροπή να λάβει μέτρα τα οποία θα συνάδουν με τα διάφορα ε, και προδιαγραφές στους οποίους θα πρέπει να υποκούν οι δικές μας επιχειρήσεις και αυτές που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείτε να έχετε ε, διαφορετικούς ε, κανόνες ε, χωρίς εσείς να εφαρμόσετε τους και να δεχθείτε ότι και εσείς πρέπει να απομειστείτε ένας μέρος της ευθύνης. Ευχαριστώ. Η Μαρία, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω παρακαλώ κάτι να γίνει με την θερμοκρασία της αίθουσας, η οποία είναι πάρα πολύ... Ε, υψηλή και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το αντέξουμε στο τέλος. Παρακαλώ να γίνει κάτι. Ναι, ναι, ναι, όντως κάνει πολύ ζέστη, όπως λέει η Μαρία Μπαθάν. Παρακαλώ λοιπόν τους αρμόδιους να ασχοληθούν με το θέμα της θερμοκρασίας. Πάρα πολύ σύντομα η Επιτροπή, ο κύριος Μπάσμανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τον εισηγητή Χαιρετίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης και τα σχόλια τα οποία ήταν, ήταν θετικά, ήταν πολύ καλή συζήτηση, σας ευχαριστούμε. Όπως ελέγχθη ήδη, το θέμα αυτό του του πληθυσμού είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει όλο και περισσότερο πρόβλημα στους πόρους τους οποίους έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι δεδομένο ότι έχουμε όλο και λιγότερο πάρό, αλλά θα πρέπει να του χρησιμοποιούμε στα πλαίσια τη πολιτική μας με τον πιο ευφυή τρόπο και θα πρέπει να κάνουμε τι σωστές πολιτικές. Επίσης, ε, υπάρχει το θέμα της ε, αηφορίας ε, της, ε, των περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η αποδοτικότητα των πόρων είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της κοινωνίας του εμπορίου και ένα από τα κύρια θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε εμείς τα πλαίσια στρατηγικής του 2020 είναι αυτό το θέμα. Θα... Αυτά ήταν τα σύντομα σχόλια που ήθελα να κάνω. Σας ευχαριστώ. Τελικές παρατηρήσεις, Σαλβατόρα Γιακολίνο. Ναι, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή τις ε, παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων. Χαιρετίζω τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλια που έγιναν όταν θα πρέπει να εν τελική έκδοση και τις προτεραιότητες του θέματος αυτού. Νομίζω ότι περισσότεροι συνάδελφοι συμμερίζονται τις απόψεις μου. Ξέρουμε ποια είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και η ψηφοφορία θα γίνει στις 28 Μαρτίου. Όπως ξέρουμε, σας ευχαριστώ. Το μεσημέρι της δοσματιλογική προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Περνούμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξης. Χαιρετίζουμε τον Πασκαλ τον καλωσορίζουμε στην συνάντησή μας. Είστε εδώ μετά από την 8η συνάντηση των Υπουργών στην ε, Γενέβη. Δεν θέλω να σας προκαλέσω. Θα ήθελα να πω ότι στην ε, Γενέβη έγιναν διάφορες συζητήσεις μετά από την τελευταία των διάφορων συζητήσεων της γύρω την Τόχα. Τι θα κάνετε και τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς ε, για να ε, μπορέσουμε να ξαναθέσουμε σε εκκίνηση όλες αυτές τις συζητήσεις. Φαίνεται ότι έχουν φτάσει σε μια στασιμότητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντα με μεγάλη ευχαρίστηση επανέρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσω βεβαίως να απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που είναι οι πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές τις οποίες διερχόμαστε ανά τον κόσμο τώρα τελευταία. Βεβαίως, με την ε, εμφάνιση πολλών νέων ε, αναδιωμένων, από χωρών που είναι σήμερα ενεργοί παίκτες στην παγκόσμια οικονομία και τους οποίους παρέχουμε αναπτυξιακή βοήθεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται και προσαρμογές στα μοντέλα ε, πάρα πολύ γρήγορης ανάπτυξης τα οποία είχαμε την τελευταία δεκαετία ή έχουμε ανάπτυξη παγκοσμίως η οποία επιβραδύνεται ε, νέες αλλαγές οι οποίες πραγματικά επηρεάζουν την ε, οικονομία, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος δεν είχε τα κατάλληλα κανονιστικά πλαίσια και γι' αυτό οδηγηθήκαμε στην κρίση του 2008. Όλες αυτές λοιπόν οι θεμελιώδεις αλλαγές έχουν αντίκτυπο στο σύστημα του ΠΟΕ. Αυτή τη στιγμή είναι στα πλαίσια του ΠΟΕ πιο ε, δυναμικοί παίκτες οι αναδυόμενες χώρες. Η νομοθετική μας λειτουργία είναι ο ένας τομέας και στα πλαίσια των συζητήσεων, στα πλαίσια της, των συζητήσεων της Δόχα, βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων δεδομένων χρόνων, ώστε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι δίκαιο. Έτσι έχουν τα πράγματα και αυτό υπάρχει ε, αυτό το πρόβλημα στις ε, διαπραγματεύσεις και γι' αυτό θα πρέπει εμείς να επανέλθουμε με προσεγγίσεις εναλλακτικέ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε θέματα που μας αφορούν. Επίσης βλέπουμε ότι ε, πάρα πολλά από τα πιο πτωχά μέλη του ΠΟΕ χρησιμοποιούν το εμπόριο σαν μέσον ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία για μας. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η παρούσα κρίση δεν μειώνει την συλλογική δέσμευση που έχουμε αναλάβει, δηλαδή να βοηθήσουμε τις πιο φτωχές χώρες να αναπτυχθούν και θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, συν τα κράτη-μέλη, ενεργούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, πράγμα το οποίο φαίνεται και στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά το εμπόριο, την ανάπτυξη και το, το εμπόριο και την ανάπτυξη. Όπως ξέρετε, και το εμπόριο αλλάζει. Γιατί? Διότι τι είναι το εμπόριο σήμερα αλυσίδες παγκόσμιες αγαθών. Δηλαδή, προστιθέμενη αξία για εισαγόμενα αγαθά, τα οποία επανεξάγονται με υψηλότερη αξία και με περισσότερη εργασία εκ μέρους κάποιων. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αναπροσαρμοστούμε αυτό, σε αυτό το γεγονός, πώς θα μπορέσουμε να μετρήσουμε ε, με άλλα μέτρα και σταθμά το εμπόριο, διότι μετρούμε τις ροές, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές, κάθε φορά που κάποια αγαθά περνάνε τα σύνορα, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ ακριβή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει ε, το εμπόριο στην ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην ανάπτυξη και στη μείωση της στόχης. Έτσι λοιπόν έχουμε μια στρεβλή εικόνα για τι ανισορροπίες που υπάρχουν και δεν μπορούμε τον 21ο αιώνα να συνεχίσουμε να μετράμε το εμπόριο με τα μέτρα και σταθμά του 19ου αιώνα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες ε, αναπροσαρμογές για να μπορέσουμε και να αλλάξουμε παραπάνω για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ε, τα πράγματα και να μετρούμε το εμπόριο ε, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό προσπαθούμε. Ε, εγώ πρέπει να πω, έχω θέσει σε κίνηση μια νέα πρωτοβουλία που λέγεται Made in the World με τη συνδρομή του ΜΑΟΣΑ, του Ιαπωνικού Τζίτρο, την Eurostat, του ITC, των ΗΠΑ, ώστε να μπορέσουμε να μετρήσουμε διαφορετικά το εμπόριο εμείς που κάνουμε την πολιτική καθώς και η επιχειρηματική κοινωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ε, μας βοηθήσει να μετρήσουμε διαφορετικά την ε, ανάπτυξη διότι αυτές οι παγκόσμιες αλυσίες μας υποχρεώνουν κατά κάποιο τρόπο να δούμε διαφορετικά και το θέμα του προστατευτισμού. Διότι πολλοί θέλουν να το παρουσιάσουν ως κάτι το πάρα πολύ αλλά ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ε, κάνει να προχωρήσουμε και ο προστατευτισμός δεν μας προστατεύει. Επίσης, τι βλέπουμε. Πάρα πολύ υψηλό αριθμό διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. Το πολυμερές εμπόριο έχει ανοίξει και συνυπάρχει με διάφορες περιφερειακές και διμερείς πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται. Αυτό το οποίο μας απασχολούσε παραδοσιακά ήταν οι δασμοί. Αλλά όλο και περισσότερες, ε, όσο περισσότερες δίτες συμφωνίες υπάρχουν, όλο περισσότερο μπορούμε να φανταστούμε ότι σιγά σιγά θα μειώνονται οι δασμοί, πράγμα το οποίο είναι θετικό. Αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε σε όλες αυτές τις νέες διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες οι οποίες ε, ε πολλαπλασιάζονται αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε και όλα τα κανονιστικά θέματα και να έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο διαφορετικά ε, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο και μπορεί να αυτό να οδηγήσει και σε αύξηση του κόστους. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα πλαίσια ε, του διεθνούς εμπορίου σήμερα, όλο και περισσότερο ε, διμερείς περιφερειακές συμφωνίες υπάρχουν, όλο και λιγότερο ε, πολυμερείς, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα κανονιστικά ε, πρέσια, δεδομένου ότι αυτός ο κατακαιρματισμός μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του παγκοσμίου συστήματος εμπορικών συμφωνιών που έχουμε και με μεγάλες προσπάθειες έχουμε προσπαθήσει να οικοδομήσουμε το 1947. Αυτό δεν είναι καλά νέα για πολλούς από μας. Οι μεγάλοι ή μικροί είμαστε. Τα μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να αρχίσουν να εξετάζουν Ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια στο εμπόριο σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς πώς θα μπορέσουμε να διαθετήσουμε τα διάφορες ανταλλαγές στο εμπόριο χωρίς να στιάζουμε αποκλειστικά την προσοχή μας στα θέματα των μη δασμολογικών Θα πρέπει να δούμε περισσότερο πώς αναπτύσσονται οι υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες σήμερα ε, ενσωματώνονται στο κόσμο κατασκευής και στο μπορεί ακόμη σε θέματα γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες και οι προδιαγραφές και κυρίως αυτοί που ισχύουν για τον ε, ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό απεφάσισα να συγκαλέσω μία διάσκεψη ε, των ενδιαφερεμένων το πάνελ των multi-stakeholders, για να δούμε ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια στο εμπόριο σήμερα. Το 2012 δεν θα πρέπει να χαθεί για τον ΠΟΕ. Έχουμε πολλά θέματα στα πλαίσια των ε, ατζέντα ε, της ΔΟΧΑ τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν, να ολοκληρωθούν διότι υπάρχουν σαφή οικονομικά ωφέλη και ε, θα πρέπει να επιτύχουν συμφωνία την διευκόλυνση του εμπολίου. Υπάρχουν λοιπόν τομείς στους οποίους θα προχωρήσουμε όπως Φερρυπίν Ε, θέματα για τη διευκόλυνση του εμπορίου, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολλές χώρες εξετάζουν το πώς θα μπορέσουν οι, με μέτρα εξισορρόπησης οι καθήμοι από αυτές να διευκολύνουν ε, το εμπόριο. Επίσης, υπάρχουν και αναμενόμενες προσχωρήσεις των ΠΟΕ από χώρες όπως η Σερβία, το ή το Λάος. Οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά και ελπίζω ότι μπορέσουν να ολοκληρωθούν ε, σύντομα. Και όπως ξέρετε υπάρχουν και θέματα εποπτείας με τα οποία ασχολούμαστε κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών κρίσης Ελπίζουμε ότι το σύστημά μας θα ενισχυθεί, όσο και αν είναι ε, καλό αυτό το σύστημα εποπτείας που έχουμε και επαγρύπνηση, θα πρέπει να το ενδυναμώσουμε και υπάρχουν βεβαίως και άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το θέμα, τα θέματα των κρατικών ε, προμηθειών και το θέμα της προσχώρησης αυτές τις ε, συμφωνίες της Κίνας, που είναι μια νέα σημαντική αναδυόμενη χώρα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα για το ε, πολυμερές εμπόριο. Δεν νομίζω ότι και μεγάλη, υπάρχει μεγάλος ε, συνδυασμός εκ μέρους των μελών μας να συνεργαστούν στα πλαίσια ενός πολυμερούς πλαισίου για να μπορέσουν να προχωρήσουν περαιτέρω στην ε, επίλυση των ε, προβλημάτων και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζει σήμερα το εμπόριο. Στα πλαίσια της οικογένειας των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών ε, δεν υπάρχει και μεγάλη βούληση να μειωθούν οι εκπομπές θερμοκηπίου. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, το σύστημα το οποίο οικοδομήσαμε με προσπάθειες εδώ και χρόνια, να συνεχίσουμε να το ενισχύουμε και όχι να το διότι αυτό το παγκόσμιο σύστημα, το εμπορικό, νομίζω ότι συνεισφέρει στην ευημερία όλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν με εκπλήσει το ότι πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε στο χρόνο που σας έχει δοθεί. Ο Κύριος Κάσπαρη από το ΕΚΔ. Ευχαριστώ κύριε Λαμή. Χαίρομαι που είστε εδώ, αλλά είναι καλό δείγμα ότι έχετε τόσο χρόνο και μας επισκέψετε. Καλύτερα να ήσασταν πολύ άσχολος και να είχατε λιγότερο χρόνο αλλά για όλα τα θέματα τα οποία αναφέρατε δύο με ενδιέφεραν περισσότερα διότι βλέπουμε ότι στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής αναμένει κανείς ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η πολιτική αυτή και άλλα θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά πρότυπα και ε, ε, ανθρώπινα δικαιώματα οπότε θα ήθελα να ξέρω πώς συνεργάζεστε με τους άλλους οργανισμούς στον τομέα αυτό, με την ΙΕΟ, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαβλέπετε στην φάση της αδρανίας των πολυμερών διαπραγματεύσεων ότι το 2012 θα μπορούσε να είναι το έτος όπου θα προχωρήσει ε, στις διαπραγματεύσεις αυτές ο ΠΟΕ ε, και ότι θα μπορέσουν να επιληθούν και άλλα θέματα όπως ο μηχανισμός επιλύσεως των διαφορών για να μπορέσει να αποδεσμευτεί ο ΠΟΕ ε, από διάφορα θέματα όσον αφορά τον προστατευτισμό το οποίο θίξατε επίσης με ανησυχεί πάρα πολύ διότι όλο και περισσότερα με κράτη-μέλη του ΠΟΕ παρουσιάζουν θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την, ε, τις αρμοδιότητες του ΠΟΕ. Ότι έκανε η Αργεντινή και η Βραζιλία. Τώρα οι Κινέζοι είπαν ότι θέλουν όλο το κράτος να κατακλειστεί με ε, αυτοκίνητα. Ε, θεωρείται ότι ο ΠΟΕ είναι αρκετά ισχυρός οργανισμός κατά τρόπο Ωστόσο λοιπόν ε, να πιέσει ε, τα κράτη-μέλη να σεβαστούν ε, τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και αρχές και επιπλέον ποια κράτη μέλη παραβιάζουν ορισμένους κανόνες του ΠΟΕ και θα πρέπει να τεθούν πρώτων ευθυνών τους το 2012 διότι εάν θέλει να επιβιώσει ένας οργανισμός πρέπει να εξελίσσεται και αυτό με ανησυχεί. Δεν θα ήθελα να αποδυναμωθεί ο ΠΟΕ. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ΠΟΕ, μία ισχυρή ένωση κρατών που έχουν ε, ένα ισχυρό πρόγραμμα και δεν θα ήθελα να αποδυναμωθεί ο οργανισμός αυτός ε, στο τρέχον έτος και ε, θα ήθελα να μας περιγράψετε τις πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να αναλάβετε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Θα σας παρακαλούσα να είστε σύντομος. Ο επόμενος είναι ο κύριος Λάνια από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά ε, και πάλι δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ότι εσείς αναφερθήκατε ε, στην παγκόσμια ρύθμιση, ενιαία ρύθμιση. Αν σκεφτώ όμως την Ιταλία ή τους εργαζομένους στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Γερμανία και να πιστεύω ότι τα προβλήματα πρέπει να επιληθούν παγκοσμίω νομίζω ότι δεν είναι πολύ πιστική αυτή η αντιμετώπιση ενώ <clears throat> με ε, διμερείς διαπραγματεύσεις μία βιομηχανία μπορεί να επιληθεί πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, εσείς πώς θα διευκολύνετε την παγκόσμια ρύθμιση των προβλημάτων. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε γι' αυτό και τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς επί του θέματος. Έχετε καταρτήσει μία ομάδα που σκέφτεται τα θέματα αυτά και θα ήθελα να μας πείτε πού έχει καταλήξει μετά από ένα τρίμηνο. Και επίσης ο κύριος Γκασπάρη αναφέρθηκε στον προστατευτισμό, τον οποίο διαπιστώνουμε σε πολλούς τομείς και οι διαδικασίες είναι πολύ μακριές, ε, μακριές για να μπορέσει να υπάρχει σωστός έλεγχος. Μπορεί ο ΠΟΕ και εδώ όντως να παρέμβει ε, πιο ε, ισχυρά για να βελτιώσει τις διαδικασίες και κατά τρόπον ώστε να αποδιώξει ο ΠΟΕ το, το, τα θέματα του προστατευτισμού που δεν έχουν καμία σχέση με το έργο του. Η Κάθριν Μπίλτερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λαμή που μας μιλήσατε. Είπατε ότι δυσκολευόμαστε να περάσουμε από τα μέσα του 19ου μετά στον 20ο και τώρα στον 21ο αιώνα. Και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς βλέπουμε εδώ πέρα τις διαφορές στο GSP. Ίσως αρχικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον συντελεστή ε, αν, ανθρώπινης ανάπτυξης αντί το, του ΑΕΠ. Υπήρξε έκθεση της Επιτροπής, θα τη διαβάσω, ενώ το HDLI είναι ε, διεθνώς αποδεκτός εντελεστής δεν είναι αποδεκτός ε, για ένα μονομερές προτιμησιακό ε, σχέδιο του ΠΟΕ. η χρήση μόνο οικονομικών κριτηρίων και ε, προτιμήσεων δεν βοηθάει πάντα. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη. Θέλετε να εξετάσετε και άλλες πληροφορίες, γιατί στη δική μας Επιτροπή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να καταστήσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις δίκαιες και βιώσιμες. Ευχαριστώ. Thank you. Now, the Ευχαριστώ, Πρασίνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, <clears throat> ευχαριστώ κύριε Λαμέ, ε, χαίρομαι που ήρθατε εδώ. Ο, μ' άρεσε η αναφορά στο Made in World και στην Γαλλία στην προεκλογική εκστρατεία θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Αλλά εδώ αναφέρεστε στην κρίση ε, του πολυμερισμού και υπάρχουν ε, περιφερειακές ομάδες και πρέπει κανείς να σκεφτεί πώς δια διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις. Αν αναστρέψουμε όμως το σκεπτικό πρέπει να δούμε ποια πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση διότι είπαμε το, ότι το πολυμερές πλαίσιο θα είναι το καλύτερο αλλά ποιο θα είναι ε, το, ποια θα είναι η προσέγγιση της Ευρώπης. Δεν σκέφτομαι εδώ μόνο αυτούς που θα σας ε, αντικαταστήσουν αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η ιδέα για τη θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο εμπόριο διότι στην αρχή υπήρχε στο πρόγραμμά σας μία ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών αλλά ε, υπήρχε και μία σκέψη για τις ρεαλιστικές διαστάσεις του εμπορίου ενώ τώρα υπάρχει ε, μία ζώνη ελευθέρων συναλλαγών η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις ε, σκέψεις και τις συζητήσεις οι οποίες υπάρχουν εντός των κρατών μελών και εδώ δεν θα ακολουθώ τον Μπέρντ Λάνιε αλλά αμφισβητούμε τις ε, δημόσιες προμήθειες διότι εάν ε, ε, αυτές οι δημόσιες προμήθειες δεν είναι ένα μέσο πολιτικής ε, βιομηχανικής, δηλαδή δεν είναι ένα μέσο σε ορισμένους τομείς που θα έπρεπε ίσως να είναι ενδιαφέρον και να προωθηθεί, διότι βλέπουμε τις συναλλαγές της Ιαπωνίας με τον Καναδά στο θέμα αυτό και μία στροφή της οικονομίας και ε, ενδιαφέρουσες ανταλλαγές οι οποίες δεν είναι υποχρετικά ενάντια στις υπόλοιπες αλλά που προωθούν και ε, την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Ε, και τέλος αναφερθήκατε στις πολυμερείς συναλλαγές. Η Ευρώπη από τον τομέα αυτό πάντοτε έχει προωθήσει και εμπορική πτυχή. Αλλά τι θα γίνει τώρα ε, στην Ευρώπη εάν εάν οι εταίροι της δεν κάνουν προσπάθειες θα πρέπει ε, να προωθήσει την αποτυχημένη πολυμερή συνεργασία σχετικά με το διοξίδιο του άνθρακος με άλλους τομείς δηλαδή μήπως πρέπει να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες εάν τις έχουν εγκαταλείψει εγκαταλείψει άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέρνη, Ευρωπαίος Συντηρητικός. Ευχαριστώ. <clears throat> Καλώς ήρθες Πασκάλ, χαίρομαι που σε βλέπω. Είχαμε τον ε, Αμερικανό προσωπευτή Πλάνκετ που μας επισκέφθηκε ε, πριν λίγο καιρό και μας α, ε, μίλησε για μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Είναι ένας όρος που αγαπούν οι Αμερικανοί και είπε στη συνέχεια ότι κατά τη γνώμη του οι πολυμερείς ε, συμφωνίες είναι μια καλή εναλλακτική ε, στην ε, μονομερή προσέγγιση που έχει τελματώσει. Ξέρουμε ότι γενικά είναι καλύτερη προσέγγιση βεβαίω η μονομερή. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη δική σα άποψη, αν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πτυχή για να επανεκκινήσουμε το παγκόσμιο εμπόριο. Γιατί υπάρχει και ε, η πλευρά του ειρηνικού εκεί πέρα και υπάρχουν διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ. Υπάρχει από την άλλη και το θέμα της Ρωσίας ε, και τις συνδέσεις με τον ΠΟΕ, υπήρξε, κάποιοι μίλησαν για θρίομβο, κάποιοι άλλοι έχουν αμφιβολίες. Πολύ συχνά ξέρουμε ότι έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας και ότι έχετε συχνά, συχνά επαφή μαζί μας. Μήπως ο ΠΟΕ θα έπρεπε να δίνει μια τήσια έκθεση, όχι μόνο για την ε, Ρωσία, αλλά για τη γενικότερη κατάσταση, για να δούμε αν ε, ακολουθούν ε, τους κανόνες του ΠΟΕ όπως εσείς ε, καθορίζετε. Και τώρα, από ό,τι έμαθα, η Ρωσία έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω παθήσεων, οι οποίες όμως μεταφέρονται μέσω παρασίτων, όχι μέσω του κρέατος. Δεν ξέρω αν έτσι συμμορφώνονται, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου και το πνεύμα της ερμηνείας. Παρακαλώ να το σχολιάσετε. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ. Εκτιμούμε που έρχεστε εδώ συχνά. Thank you, Ευχαριστώ. Helmut Scholz από την ΚΟΕ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι ήρθατε να επισκεφτείτε την Επιτροπή μας και νομίζω ότι εδώ το σύνθημα το οποίο ε, ε, συγκεντρώνει τις ε, περισσότερες απόψεις είναι ο πολυμερισμός και ιδίως στις υποανάπτυξη χώρες και στις αναδιόμενες χώρες ελπίζει κανείς ότι ο ΠΟΕ θα διατυπώσει μία νέα μορφή του πολυμερισμού που θα εφαρμοστεί στον 21ο αιώνα. Ο ΠΟΕ λοιπόν δεν θα έπρεπε να μπορέσει να προωθήσει κάτι το οποίο νόμος θα αμφισβητήσει μακροπρόθεσμα τον ρόλο που διαδραματίζει διότι με την συμμετοχή ε, της ε, Κίνας ιδίως ε, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε 4 δισεκατομμύρια μεταξύ Κίνας και Ινδίας με 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους που αποτελούν μέρος της πρέπει να σκεφτούμε πώς θα έχουν πρόσβαση στους σπόρους, πώς θα τραφούν και αυτά είναι τα τέσσερα δέκατα του πληθυσμού της εμφυλίους. Χωρίς να σκεφτώ τα άλλα τρία δέκατα που είναι η Αφρική και οι ε, ε, υποανάπτυξη χώρες. Πώς θα υπάρχει δηλαδή ε, μία σύγχρονη ανάπτυξη και πώς θα υπάρχει υπάρξει ένα νέο προφίλ αυτού του οργανισμού διότι αναρωτιέμαι εάν υπάρχει κάποια σκέψη για τέτοιες εξελίξεις στον ΠΟΕ ε, υπάρχουν και τα σχόλια της Βραζιλίας στην διακυβερνητική διάσκεψη ε, σχετικά με τον οργανισμό που χρειάζεται για τις υπηρεσίες και προτείνεται ε, τι γίνεται, τι θα γίνει με την ε, γεωργία, πώς ε, θα ε, απελευθερωθεί η γεωργία και αυτό το θεωρώ ότι είναι μία αντίφαση με το παρελθόν σας σαν επίτροπος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κερδοσκοπία, γνωρίζουμε ότι υπάρχει προβλήματα και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Κασπάρη πώς δηλαδή θα μπορέσει ο ΠΟΕ να κάνει τα βήματα που χρειάζεται για να μπορέσει να εξελιχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας δώσουμε το λόγο σε άλλα μέλη της Επιτροπής. Από εδώ και πέρα έχετε 1,5 λεπτό για τις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με τη Λουσία Αντρικένα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Λαμή. Αζερβαϊτζάν και Κίνα. Το Αζερβαϊτζάν προσπαθεί να γίνει μέλος ε, του ΠΟΕ από το 1997. Έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος. Έχουμε βρεθεί σε αξία αδιέξοδο. Ποιε είναι οι αιτίε ε, για αυτό το... αυτή την κατάσταση κατά τη γνώμη σα και τι πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον. Και πάλι Κίνα και ΠΟΕ, ε, ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση. Ε, και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την ε, κατάσταση. Κατανοούμε ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις και πάλι θα ήθελα να, μας, ε, να ακούσω τη δική σας εκτίμηση. Ευχαριστώ. Your Grastrix από S&D. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω ουσιαστικά δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, έχω την εντύπωση ότι ο ΠΟΕ ε, στο φόσο των διαπραγματεύσεων της Ντόχα δεν έχει πετύχει και πολλά και αυτή είναι η γενική εντύπωση την οποία αποκομίζουμε. Μπορεί ίσως να σκεφτεί κανείς ότι ίσως και η οργανωτική δρομή του ΠΟΕ ε, ε, ευθύνεται για αυτή την αποτυχία ε, και για το ότι δεν υπάρχουν θεαματικές εξελίξεις τον τελευταίο καιρό ε, και ε, υπάρχει καμία συζήτηση για το μέγεθος του ΠΟΕ αν ε, ε, πρέπει στο μέλλον να συμμετέχουν τα κοινοβούλια ή όχι είναι κάτι το οποίο σκέφτεστε προβλέπετε ε, καμία αλλαγή στη δομή του οργανισμού στο μέλλον και ο συνάδελφος κύριος Σόλτς μας είπε ότι συζητάμε μια πολυμερή συμφωνία όπως τη συμφωνία συμφωνία άκτα η οποία είναι πολύ αμφιλεγόμενη από πλευράς περιεχομένου αλλά ε, αυτή η συμφωνία συνήφθη εκτός του ΠΟΕ και ε, όσον αφορά την άποψη των πολυμερών συμφωνιών την οποία εμείς πρεσβεύουμε αυτό δεν ακολουθεί καθόλου αυτό το σκεπτικό. Η κυρία Μπαντία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε κύριε Λαμή την παρουσία σας εδώ σήμερα. Οι παρεμβάσεις σας και οι συναντήσεις που οργανώνετε πάντα είναι πολύ επικοινωνικές αλλά μας ανησυχούν. Μας μιλάτε για αυτή την ε, νέα όψη του παγκοσμίου εμπορίου, για τις αλλαγές που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία και των κυβερνήσεων και των επιχειρηματιών και όλων των φορέων. Δεν θα σας κάνω μία απευθείας ερώτηση, αλλά θα σας ερωτήσω το εξής. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να λέμε στους παραγωγούς και στους επιχειρηματίες Ευρωπαίους αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις ίδιες ιδέες που χρησιμοποιήσαμε τώρα, δεδομένου ότι έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές. Τι πρέπει να τους πούμε ότι πρέπει να κάνουν, δηλαδή ότι μακροπρόθεσμα ε, θα πρέπει να έχουν καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη κατάρτιση, αλλά θα πρέπει να το ρίξουν στις εξαγωγές, δεδομένου ότι έρχεται τόσο μεγάλη κρίση Ευρωπαϊκή Τι θα πρέπει να τους πούμε. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ζωζέφ Ανδρέας. ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λαμή για την παρουσία σας εδώ και διότι προσπαθείτε να μας εξηγήσετε πώς έχουν τα πράγματα στον τομέα του εμπορίου του οποίου το πρόσωπο αλλάζει. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ω ε, εισηγήτρια για την μεταρρύθμιση αλληλευτική ε, πολιτική, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι για τα τα θέματα τη αλληλείας σε κάποιες χώρες, δεδομένου ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά πάρα πολύ και κυρίω τι γίνεται με την Ιαπωνία, την ε, Κίνα και τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Λαμή και σας ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέτετε παρόλο που όπως είπε και ο κύριος Γασπάρη θα προτιμούσαμε να σας δούμε στην διαπραγματεύσει και όχι εδώ. Για τον ΠΟΕ. Αν ισχύει αυτό που μου λένε πολλοί συνάδελφοι και πολιτικοί ότι πράγματι μας αρέσει ε, ο πολυμερισμός, αυτό είναι ε, το καλύτερο αλλά δεν λειτουργεί, γι' αυτό πάμε σε διμερείς σχέσεις. Ναι, αλλά αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Μήπω πρέπει να το δούμε από το ή κλαδική άποψη. Γιατί βλέπουμε συχνά στον ΠΟΕ ότι ε, η γεωργία ε, κρατά τι ε, διαπραγματεύσει και στους άλλους τομείς, όπως, ας πούμε στη βιομηχανία. Και μετά με τη σειρά του κρατά τι διαπραγματεύσει στις υπηρεσίες υπάρχουν χώρε όπου ε, οι υπηρεσίε αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του ΑΕΠ. Και αν ε, καταφέρουμε να έχουμε καλύτερε διαπραγματεύσει, τότε θα δημιουργήσουμε καλύτερε συνθήκε σε όλο τον κόσμο. Παζαλεύσκη είναι ο τελευταίο ομιλητή από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Γενική Διευθυντή, έχω ένα σύντομο ερώτημα. για την εγκαθίδρυση της Τελωνιακή Ένωσης ε, Ρωσίας, ε, Καζακστάν ε, και άλλων. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος για την εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ δεδομένης αυτής της Θελωνακής Ένωσης μεταξύ Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζακστάν. Καθότι δεν είναι όλες αυτές οι χώρες μέλη του ΠΟΕ ενδεχομένως να μπορέσουν να ε, παρακάμψουν τους κανόνες του ΠΟΕ. Και δεύτερον, θεωρείτε ότι θα μπορούσε και η Λευκορωσία να γίνει μέλος ε, του ΠΟΕ. Πασκαλαμή. Ακούστηκαν πολλά ερωτήματα. Έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε. Θα τα πάρουμε τη σειρά. Για το ερώτημα του κύριου Κασπάρη. για την πειθαρχική προσέγγιση, τη συνεργασία με άλλες νησίδες ε, στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Ναι, αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου και με τον ILO και με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, ε, με, τον οργανισ... με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, με το ε, Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων. Υπάρχουν τώρα δύο ε, με όλους αυτούς τους οργανισμούς Κάποιες φορές έχουμε καταλήξει και σε κοινέ ε, εκθέσεις ή ανακοινώσεις ε, με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για το περιβάλλον ε, και τη διατροφή. Συμμετέχουμε ιδιαίτερα ενεργά στην Task Force για την Επιστημική Ασφάλεια που συστάθηκε την περίοδο της κρίσης. Υπάρχουν λοιπόν γέφυρες συνεργασίας όμως πράγματι όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν ε, δικά τους ε, καθήκοντα, δικές τους αρμοδιότητες ε, και λαμβάνουν οδηγίες από τα μέλη τους. Εφόσον η σκέψη ότι επειδή όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν τα ίδια μέλη, άρα είναι δεδομένη και στην εργασία, είναι λογική αυτή η άποψη, αλλά από πρακτική άποψη δεν ισχύει υπάρχουν μέλη αυτών των ε, οργανώσεων που αποφασίζουν εάν πρέπει να υπάρξει συνεργασία ή όχι. Εμείς ως ε, γενικοί διευθυντές, οι γενικοί γραμματείς έχουμε ένα περιθώριο λεγμών, αλλά εάν ας πούμε μέλη της Διεθνής Οργάνωσης της Εργασίας δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη εντολή που δίνει τη δυνατότητα ε, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασία να έχει καθεστώ παρατηρητή ε, στον ΠΟΕ, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τώρα, το γεγονό ότι είναι τα ίδια μέλη και στον ΠΟΕ και στον ILO, κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια και καθεστώ παρατηρητή. Αλλά Απλώ μέλη της Διεθνής Οργάνωσης εργασία δεν έχουν πάρει τέτοια απόφαση. Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν περιορισμοί σε αυτή τη συνεργασία. Και τα μέλη ε, αποφασίζουν ποιοι θα είναι αυτοί οι περιορισμοί. Τώρα για τον προστατευτισμό, τεράστιο ζήτημα. Υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα που ορισμένες φορές θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Πρώτον, υπάρχουν διεθνείς ε, κανόνες που πρέπει να τηρούν ε, οι χώρες. Δεύτερον, τους σέβονται αυτούς τους κανόνες οι χώρες. Ας μην ξεχνούμε όμως το πρώτο ερώτημα. Υπάρχουν πολλοί τομείς ε, της εμπορικής και εποχηματικής ζωής που δεν ρυθμίζονται από διεθνείς κανόνες. Δεν υπάρχει συμφωνία του ΠΟ, για παράδειγμα, για τη διαφθορά. Παρότι γνωρίζουμε ότι η διαφθορά αποτελεί ε, πρόβλημα ε, στην επιχειρηματική ζωή πολλών χωρών ε, του κόσμου. Υπάρχουν κανόνες δασμολογικοί για τις δημόσιες επενδύσεις, παρόλο που δεν είναι κανόνες του ΠΟΕ, είναι διμερείς. Επομένως, εάν η άποψη είναι ότι κάποιες από αυτές τις πρακτικές θα πρέπει να ρυθμίζονται από διεθνείς κανόνες, ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι μέσω ε, κυρίαρχων κρατών που θα πρέπει να αποφασίσουν ότι πρώτον υιοθετούν εντολή διαπραγματεύσεων αυτών των κανόνων και δεύτερον ότι θα επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις. Μετά υπάρχει και άλλο ερώτημα όταν υφίστανται κανόνες γίνονται σεβαστοί. Και βεβαίως εδώ ο ΠΟΕ είναι ιδιαίτερα ισχυρός οργανισμός. Είναι ο μοναδικός οργανισμός όπου οι διεθνείς ε, κανόνες ε, συνεχώς ε, την χάνουν εξέτασης, αναθεώρησης, παρακολούθησης. Και στο δικό μας σύστημα, εάν συμμετέχει στη διαδικασία, οφείλει να ε, συμμορφωθεί με τους ε, κανόνες του ΠΟΕ. Επομένως, έχει μια μεμονωμένη χώρα το δικαίωμα να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πρώτον, κοιτάζουμε αν υπάρχει κανόνας και δεύτερον, αυτός ο κανόνας σίγουρα θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Για παράδειγμα, έχουμε την Κίνα. Η Κίνα τηρεί τις δεσμεύσεις της. Ναι, τη τηρεί. Εάν όχι, εάν δεν τη στηρίσει, οποιοδήποτε κράτος ε, μέλος ε, του ΠΟΕ μπορεί να οδηγήσει ε, την ε, Κίνα σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών και η Κίνα έχει κερδίσει τις μισές υποθέσεις και έχει χάσει τις άλλες μισές. Κύριε Λάγκε. Εάν οι διμερείς συμφωνίες είναι πιο αποδοτικές από τις ε, πολυμερείς, ρωτήσατε. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ποιο είναι το ποσοστό του παγκοσμίου εμπορίου που διεξάγεται σύμφωνα με διμερείς ε, συμφωνίες. 15% είναι η απάντηση. Το 85% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται υπό πολυμερείς συμφωνίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διμερείς συμφωνίες αποτελούν το 15% του παγκόσμιου εμπορίου θεωρητικά, αλλά λόγω της πολυπλοκότητας των διμερών ε, συμφωνιών ε, χρησιμοποιούνται εν μέρη μόνο από τους ε, οικονομικούς φορείς για τα κριτήρια αποδοτικότητας. Αν δηλαδή αξίζει τον κόπο να, ε, να, ξοδεύουμε τόσο χρόνο και χρήμα, αν θέλετε, για κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται πλήρως. Η δική μου ομάδα ενδιαφερομένων μερών εστιάζει την προσοχή της κυρίως ε, στο να δώσει απαντήσεις ε, στο δικό σας ερώτημα, κύριε Λάγκε. Δηλαδή, ποια είναι τα εμπόδια ε, σήμερα και στο μέλλον για το εμπόριο. Υπάρχει μια ατζέντα διαπραγματεύσεων, η αποστολή του ΠΟΕ είναι, ένα, ε, είναι το άνοιγμα του εμπορίου και αυτό σημαίνει επίλυση των ε, πραγματικών προβλημάτων και των πραγματικών εμποδίων που υφίστανται. Αυτή είναι μια διαδικασία που εγώ θέλω να ξεκινήσω. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε αυτή την ε, ομάδα. Και θα αναγγείλω την ε, σύνθεσή της ε, πολύ σύντομα. Κυρία Μπέρντα, για το GSP. Όπως ξέρετε υπάρχουν τρεις τρόποι ρύθμισης του εμπορίου, μονομερός, διμερός και πολυμερός. Το GSP είναι μονομερής προσέγγιση ρύθμισης του εμπορίου όπου εσείς και κάποιος άλλος, ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ε, ε, ε, προσφέρετε συγκεκριμένες προτιμήσεις σε ορισμένες χώρες που τηρούν συγκεκριμένους όρους που έχουν αποφασίσει να επιβάλλουν η ΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη αγορά. Ποιο είναι το κριτήριο εδώ. Έχουμε έναν κανόνα στον, ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου που έχει ελεγχθεί από την ε, νομολογία και εντάξει σε γενικέ γραμμέ, μην τα πάρετε κατά λέξη αυτά που λέω, γιατί οι νομικοί μου σίγουρα θα έχουν πρόβλημα με κάτι που δεν έχουν γράψει οι ίδιοι εδώ. Επομένω, ε, κατά προσέγγιση τα λέω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο κριτήριο θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ε, εφόσον τα κριτήρια αυτά να είναι ξεκάθαρα, αντικειμενικά και διαφανή. Αυτό αποφάσισε ε, και η αρμόδια αρχή σε μια υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Επίτροπο Νοέλ, όταν ε, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε κατά την άποψη της Ινδίας διάκριση κατά της Ινδίας. Υπάρχει λοιπόν ομολογία. Εφόσον δεν υπάρχει υποψία προτίμησης ε, συγκεκριμένων φορέων, ε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Για τον κύριο Ζαντό, ως συνήθως ε, πάτε αρκετά γρήγορα. και λέτε, χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένο το, ε, το, μονομερές ε, σύστημα το οποίο υπάρχει εδώ για 60 χρόνια. Υφίσταται αυτό το κείμενο, το, το, το σύστημα εφαρμόζεται. Βεβαίω τώρα έχουμε και μία διαμεσολάβηση την οποία δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ε, Ω ε, αποτυχημένοι και βλέπουμε όλοι στον επιχειρηματικό κόσμο όπου οι διαπραγματεύσει απλώς ε, δεν ε, προχωρούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, γενικώ είναι αποτυχημένο το σύστημα. Αυτό που ρυθμίζει καλύτερα αυτή τη στιγμή τις διεθνείς πολυμερείς σχέσεις είναι αυτό το σύστημα. Διεθνείς εμπορικές σχέσεις, νόμι, είναι το μονομερές σύστημα. Τώρα, αυτό που είπατε ότι είπα και εκείνα, δεν μπορούν να συμφωνήσουν ακριβώς τι πρέπει να ισχύει για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ναι, πράγματι υπάρχουν δυνατότητες ε, ε, προόδου, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει εξετάζοντας τα θέματα ένα προς ένα. Τώρα, για το αν ε, η αγορά του δημοσίου Συγγνώμη, αν οι κρατικέ προμήθειε μπορεί να αποτελέσει ένα τομέα, βεβαίω. Πρέπει όμω αμοιβαία να αποδεχθούμε ότι θα ανοίξουμε κάποια τμήματα των κρατικών προμηθειών. Η δυνατότητα ρύθμισης των κρατικών προμηθειών παραμένει για όλα τα μέλη του ΠΟΕ μέχρι τη στιγμή που δέχονται άλλους όρους σε αντίθεση με τους ε, όρους που αποδέχονται ε, τα άλλα συμβαλόμενα μέρη. Παραμένουν ε, ιδιαίτερα σημαντικά περιθώρια λιγμών και πάλι το, το μέλος του ΠΟΕ αποφασίζει αν, είναι, αν το συμφέρει να μπει σε, αυτή την ομάδα των χωρών που έχουν ανοίξει τις κρατικές προμήθειες σε ορισμένους τομείς με, σε ορισμένο ποσοστό για ορισμένους τομείς και όχι για άλλους. Και βεβαίω, ε, αν ανοίξει η Κίνα 20-30% τις κρατικές προμήθειες αυτό θα θα δημιουργούσε έναν τεράστιο κύκλο εργασιών ε, ε, και επενδύσεων 100-200 ε, δις κάθε χρόνο. Τώρα, κύριε Ζαντώ, εσείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να εξετάσετε το εξή θέμα. Εγώ πολύ συχνά εξετάζω του σύνεγγυς ε, τα στοιχεία που αφορούν το ευρωπαϊκό εμπόριο και ε, η, το, το η περιεκτικότητα των ε, εμπορικών συναλλαγών των ευρωπαϊκών σε, σε, άνθρακα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες. περιεκτικότητα σε διευσίδιο του άνθρακα. Και πρέπει να δείτε τι θα κάνετε σε αυτόν τον τομέα. Γιατί από περιβαλλοντική ε, άποψη θα πρέπει αυτό να σημάνει ότι η Ευρώπη θα μειώσει τις εξαγωγές και θα αυξήσει τις εξαγωγές. Το οποίο θα μας γυρίσει στο μεσαίωνα και δεν είναι ε, βεβαίως ε, αυτός ο στόχος. Αυτό βεβαίως θα το εξετάσω πολύ προσεκτικά. Κύριε Στέρντι. Τα πάντα εξαρτάται από το τι επιθυμείτε. Αν δηλαδή μια πολυμερή συμφωνία μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερε εξελίξει, ναι, αλλά υπό συγκεκριμένου όρους. Πάρτε για παράδειγμα τις υπηρεσίες. Η συμφωνία του ΠΟΕ για το άνοιγμα των ε, υπηρεσιών πάντα γίνεται Ε, το μελβερών. Όταν φτάνουμε στην αυτή την κρίσιμη μάζα του 85% ανοίγει και για τα υπόλοιπα μέλη. Αυτή είναι μία εκδοχή που συμβάλλει στο άνοιγμα των πολυμερών συμφωνιών. Τώρα, αν μιλάμε για ένα πρότυπο ε, που συνάδει με τον ΟΣΑ, το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποιο όφελος. που να συγκρίνεται με το άνοιγμα των χωρών του ΩΣΑ μεταξύ τους. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα, θα ωφελούσε και τους ε, εμπορικούς εταίρους και αυτές τις χώρες, αλλά κυρίως τις, ανα, τις αναδυόμενες οικονομίες. Και εκεί επανερχόμαστε στο ζήτημα ΙΠΑ-Κίνας. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος ε, που ε, έχουμε φτάσει σε διέξοδο. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Για τη Ρωσία, σε τη φορά την ε, ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, δεν υπάρχει κάτι σαν αυτό που υπήρχε με την Κίνα, όταν υπήρξε ένταξη της Κίνας, δηλαδή ετήσια έκθεση για την εφαρμογή. Η Ρωσία πρέπει να υποβάλει το εμπορικό της καθεστώς στα μέλη του ΠΟΕ μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Αυτή είναι η δεσμευσή τους. Και εκεί βεβαίως ε, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να θίξει οποιοδήποτε ερώτημα για το εμπορικό καθεστώς της Ρωσίας. Κύριε Σόλτς. Πολύ σημαντικό το ερώτημά σας, ερώτημά σας για το μέλλον των ε, πολυμερών ε, συμφωνιών. Κάποιες φορές έχω την εντύπωση ότι όλοι θεωρούν, ως απο... θεωρούν αποτυχία τις ε, πολυμερές συμφωνίες και ότι θα πρέπει να, να ακολουθήσουμε κάποια άλλη προσέγγιση. Αυτό άκουσα και σήμερα. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό το καθεστώς η προσέγγιση δηλαδή των πολυμερών συμφωνιών, το οποίο ακολουθήθηκε εδώ και πολλά χρόνια, δεν ήταν και πολύ πολυμερή. Πρέπει να γίνουμε πραγματικά πολυμερεί. Αν σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ ηγούνται του πολυμερού συστήματος, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μετατρέψουμε το ε, σύστημά μας όπου λόγο θα έχουν και η Κίνα και η Ινδία και η Ινδονησία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν ένα μου συμφέρον να μοιραστούν αυτό τον ηγετικό ρόλο μαζί μας. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Και αυτό σημαίνει αλλαγές ε, στην μακροοικονομική συνεργασία, στα πνευματικά δικαιώματα, παντού. Πρέπει λοιπόν να βρούμε αυτή τη νέα ισορροπία. Έχει αλλάξει ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουμε και τους κανόνες λοιπόν. Και πάλι πιστεύω ότι αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Και οι διμερείς συμφωνίες έχουν βρει κάποιους τρόπους να ξεφύγουν από αυτά τα προβλήματα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις χωρίς πολιτικές απαντήσεις στο πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή, ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ε, χωρών με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Εφόσον γνωρίζουμε ότι δεν βρισκόμαστε σε έναν ε, ασπρόμαυρο κόσμο που ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατές και ποιες είναι οι αδύναμες χώρες. Έχουν αλλάξει λοιπόν τα πράγματα και όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε. για το Αζερβαϊτζάν. Βεβαίω, η διαδικασία διαπραγματεύσεων είναι μακρά και ε, η ταχύτητα ε, εξαρτάται και από την, ε, το σκηνικό, το, σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Έχω την αίσθηση ότι η προοπτική ένταξη του Αζερβαϊτζάν υφίσταται αλλά όχι βραχυπρόθεσμα. Όπως είπα και για την Κίνα, ανέλαβε δεσμεύσεις σε πολύ συγκεκριμένε ε, τότε για μια αναπτυσσόμενη χώρα που ξεπερνούν ε, όσα είχαν δεσμευτεί να κάνουν άλλες αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Βραζιλία και άλλες. Και σε γενικές γραμμές σεβάστηκε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. Παρόλο που οι κανόνες του ΠΟΕ δεν κάλυπταν όλες τις πρακτικές σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Κύριε Δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δικαιώματα ψήφου υπάρχει πολιτικό θέμα το οποίο δεν μπορούμε να λύσουμε με το να αλλάξουμε τον τρόπο ψηφοφορίας. Έτσι και δεν έχουμε ε, ε πλειοψηφία, δεν δηλωτικούμε πλειοψηφικά στον ΕΠΟΕ, πάμε με συνένεση. Και οτιδήποτε άλλο θα δημιουργούσε μεγάλα πολιτικά προβλήματα. Το ξέρετε κι εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας πήρε 50 χρόνια να καταλήξετε σε σύστημα διπλής πλειοψηφίας. Και πάλι όμως αυτό το σύστημα δεν ισχύει για όλες τις δραστηριότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι θέμα διαδικασίας, αλλά πολιτικής. Είναι θέμα χωρών που ε, συνάπτουν μια συμφωνία που πρέπει να εγκρίνουν μέσω του κοινοβουλίου τους. Και αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Οι συμφωνίες του ΠΟΕ είναι διεθνείς συμβάσεις και αυτές πρέπει να κυρωθούν από, ε, μέσω των χώρων διαδικασιών. Για την άκτα εκτός ε, ΠΟΕ. Δεν μπορώ να σχολιάσω. γιατί παρόλο που δεν έχει υπάρξει ακόμα συζήτηση, ενδεχομένως, στον ΠΟΕ ενδεχομένως να υπάρχουν ζητήματα για την άκτα και τη συμφωνία TRIPS, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και πρέπει να παραμείνω ουδέτερος για την κυρία Μπαντιγιά. Το μήνυμα για τους Ευρωπαίους ε, επιχειρηματίες Εσείς οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες έχετε μια εξαιρετική δυναμικότητα και δυνατότητα ανάπτυξη του σημερινό κόσμο. Ποια είναι η απόδειξη το ότι κάποιοι από εσάς το κάνουν με εξαιρετικό τρόπο, άλλοι λιγότερο καλά, αλλά γιατί αυτοί οι οποίοι μεταξύ μόν που υποφελούνται πλήρως από αυτή την ανάπτυξη κυρίως των επισωμένων χωρών επιτυγχάνουν. Διότι είναι παρόντες στην αγορά με τεχνογνωσία, με μέθοδο, με προϊόντα, πράγμα τα οποία συνεισφέρει εξαιρετικά στην ανάπτυξη των, ε, του μεριδίου της αγοράς το οποίο κατέχουν παντοκοσμίου και στην ανταγωνιστικότητά τους. Και στην περίπτωση της Ευρώπης το κύριο θέμα δεν βρίσκεται στην ανταγωνιστικότητα όσον αφορά την τιμή. Δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει εμπορική και βιομηχανική ε, πολιτική ανταγωνιζόμενη το επίπεδο μισθών, αλλά πρέπει να πω ότι οι πιο ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι αυτές που βρίσκονται των θυμών και νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορεί να γίνει στην Ευρώπη είναι η ποιότητα των προϊόντων. Κυρία Ανδρέας Μπαρία, για τις ε, ε, διαπραγματεύσεις στον αλληλευτικό τομέα. Τα πράγματα προς το παρόν έχουν μπλοκαριστεί όσον αφορά τις ε, επιδοτήσεις. Έχουμε δύο διαφορετικά στρατόπεδα για αυτό το θέμα αυτό. Ξέρετε πώς έχει η συζήτηση και στην ΟΠΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τους φίλους των ε, ψαριών και τους φίλους των ψαράδων. Πράγμα το οποίο υπάρχει σε δύο στρατόπεδα και σε επίπεδο ΠΟΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα είχε αποφύγει στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων να πει αν μας είναι φίλος των ψαριών ή των ψαράδων. Κυρία Κανάλ, τομεακή προσέγγιση είναι μία από τις δυνατότητες ενδεχομένως όσων βεβαίως μπορεί να μας οδηγήσει σε μία ισορροπία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την διευκόλυνση του εμπορίου που θέλουμε. Αλλά ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με τις διαπραγματεύσεις και τομιακά. Πολλές φορές αυτή η προσέγγιση δουλεύει, πολλές φορές όχι. Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι να ρυθμίζουμε τα πάντα. Προσπαθούμε να ε, εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες, πράγμα το οποίο γίνεται και στον τομέα των υπηρεσιών από διάφορες χώρες. Πρόκειται για μία από τις δυνατότητες στις ε, διάφορες διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει τη συμφωνία στον τομέα των επικοινωνιών είχαν χρησιμοποιηθεί τέτοιες πρωτογίες, αλλά δεν κερδίζει παντής κάτω. Τώρα όσον αφορά τη Ρωσία, τον Μπελαρούς και το Καζακστάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία το Καζακστάν, το Κυρδιγιστάν ίσως. Θα προσχωρήσουν χωριστά η καθεμία. Τα μέλη της Τελωνικής Ένωσης είναι αυτά τα οποία καθορίζουν εν μέν και την εμπορική πολιτική αυτών των χωρών. Ενώ ένα άλλο μέρος είναι, ε, παραμένει στον εθνικό τομέα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά το εμπόριο. Άρα τα μέλη της ελληνικής Ένωσης προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο καθένα να ρυθμίσουν την κατάσταση ανάλογα με τα προβλήματα που έχουν ώστε να μπορέσουν σε αυτά τα δύο επίπεδα να βρουν την ισορροπία. Και συνήθως αυτό το οποίο γίνεται είναι τελωνιακή ένωση πράγμα το οποίο σημαίνει ένα συν για τον Τώρα να αφορά την Μπελάρου, Λευκορωσία. Βρίσκεται στη διαδικασία προσχώρησης και η απάντησή μου είναι παρεμφερής με αυτή την οποία έδωσα και για το Αζερβαϊτζάν. Ακόμη θα χρειαστούμε χρόνο πριν να καταλήξουμε σε συμφωνία την προσχώρηση. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος συνάντησής μας με τον Πασκάλ Λαμή. Εύκολα μπορεί κανείς να κατανοήσει γιατί ποτέ δεν μας απαγοητεύουν οι επισκέψεις του. Σας ευχαριστούμε για τις σαφείς σας απόψεις και για το ότι δεν αποκρύπτεται ποτέ την πραγματικότητα και τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Uh, Έχουμε ακόμη λίγα λεπτά μέχρι τη συνάντηση των συντονιστών και θα γίνει μία κοινή συζήτηση για δύο θέματα τα οποία είναι ε, συγγενή με τον ίδιο εισηγητή σχετικά με την Εθελοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως κεντροαφρικανικής δημοκρασίας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας στη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στη δεύτερη ε, ε, έκθεση πρόκειται για την δημοκρατία της Λιβερίας με το ίδιο θέμα έχουμε μία εξέταση αυτών των σχεδίων συμφωνίας με εισηγήτρια την κυρία Ελίζαμπετ Κιώστιγκερ από το ΕΛΚ Σα σας, έψαχνα, σας έψαχνα πιο στο πλάι, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω η συζήτηση να γίνει από κοινού και για τις δύο εκθέσεις διότι ουσιαστικά επιζητούν τον ίδιο στόχο και έχουν και την ίδια ουσία. Οπότε νομίζω ότι είναι λογικό να τα συνοψίσουμε. Γενικά θα ήθελα να πω όσον αφορά αυτές τις συμφωνίες οι οποίες έχουν σαν σύνμηση τον όρο FLECT και προσπαθούμε ε, να ε, επικεντρώσουμε τις διαπραγματεύσεις επί ενός θέματος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ενός κράτους και εδώ προσπαθούμε να περιορίσουμε την παρανομία καθότι υπάρχει τεράστια παρανομία ε, στο εμπόριο ξύλου και προϊόντος ξυλίας και και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας τεράστιος εισαγωγέας ξυλίας και προϊόντων σχετικών ε, σε ύψος 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία βιώσιμη εκμετάλλευση η οποία να επιτρέψει να ε, προωθηθεί αυτό το εμπόριο. Γι' αυτό και το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο ε, θα θέσπιζε αυτό το μέτρο του FLECT και ε, προσπαθούσε να ενισχύσει την δασική πολιτική των κρατών ε, ε, που συμμετείχαν σε αυτές τις συμφωνίες μέσω μίας σωστής πολιτικής και επιτρέποντας εισαγωγές μόνο ξυλίας η οποία θα είχε εξηλευθεί νομίμως και ε, τα μέτρα αυτά περιείχαν και χρηματοδοτικά μέτρα ε, και συμφωνίες ε, εθελοντικής συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες χώρες για να υπάρχει ένα σύστημα περί, ένα σύστημα πιστοποιήσεως της νόμιμης ξυλεύσεως των προϊόντων που που εμπλέκονται ε, και τώρα υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες και με το Βιετνάμ και επιζήτηση να υπάρξουν και διαπραγματεύσεις ε, με την Νότια Αμερική. Μέχρι στιγμής όμως τέτοιες δεν έχουν ξεκινήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2010 ασχολήθηκε με το θέμα αυτό των εθελοντικών συμφωνιών με το Καμερούν και τώρα ασχολείται ε, με την κεντρική αυτική μετά από το Καμερούν, το Κονγκό και την Κάνα κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μία συμφωνία εθελοντικής συνεργασίας να μπορέσουν να συγκεντρωθούν γύρω από το τραπέζι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ε, από το δημόσιο τομέα, από την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα της ε, εμπλεκόμενης χώρας και οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν και στη διαδικασία εφαρμογής, δηλαδή να υπάρχει μία συμμετοχή όλων σε αυτή τη διαδικασία. Στο παράδειγμα της κεντρικής αυτικής διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ακόμη αδυναμίες και η εφαρμογή χρειάζεται χρόνο μόνο όταν δηλαδή δεν θα μπορεί κανείς να ε, καταφύγει ε, σε διαφορετικές δομές για, κατά τρόπον ώστε οι συμφωνίες εθελοντικής συνεργασίας με τις χώρες της ε, Αφρικής να καταλήξει σε μια πιο αποτελεσματική πολιτική και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των χωρών που μας ενδιαφέρουν επί του προκειμένου της ε, ε, δημοκρατικής ε, ε, ε, της δημοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής και της Λιβερίας. Ε, επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ενισχύσει την αρχή της συνάψεως αυτών των συμφωνιών εθελοντικής συνεργασίας που θα πρέπει να εδρεωθούν και στο εθνικό δίκαιο των εμπλεκομένων χωρών κατά τρόπον ώστε να βελτιωθεί η δασική πολιτική και η ξύλευση στις χώρες αυτές. Ε, χρειάζονται βέβαια ενισχύσεις και ε, γι' αυτό ε, δεν θα ήθελα να υπάρχει στήριξη από τις χώρες σαν την Κεντρική Αφρική αλλά να υπάρχει μία μία πιστοποίηση ότι η κοπή της ξυλίας αυτής ήταν νόμιμη και εδώ πρέπει να παραπέμψω σε ορισμένα θέματα τα οποία ε, τονίζουν και σημειώνουν την σημασία αυτών των συμφωνιών. Δηλαδή, στη συμφωνία με την Κεντρική Αφρική ε, τονίζουμε την ε, αποτελεσματική εφαρμογή, την, ε, την συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων και την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης. Και τέλος πρέπει να μπορούν να ανατεθούν άδειες φλεκτ και είμαστε επίσης επιφυγή όσον αφορά την χρήση ε, ιδιωτικών πιστοποιητικών για την ε, ε, κοπή ξυλίας στις οποίες είμαστε αρνητικοί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο Ντέιβιτ Μάρτιν είναι ο πρώτος ο οποίος έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαν σκιώδης εισηγητής πρέπει να σας πω ότι χαιρετίζω την έκθεση και τα, την παρουσίαση που μόλις είχαμε διότι μας ενδιαφέρει το Κονγό, το Καμερούν ε, και γενικώ ε, ε, κατόπιν αυτών των συμφωνιών ε, θα πρέπει να εξετάσουμε μία προς μία και τις επόμενες συμφωνίες όσον αφορά την Κεντρική Αφρική με απασχολούν οι ηθαγενείς της χώρας αυτής διότι δεν θέλουμε να υπάρχει μια εκμετάλλευση του ε, βροχοδάσους εις ε, την περιοχή αυτή και ελπίζω των τροπικών δασών στις περιοχές αυτές και θα ήθελα να τονιστεί το θέμα και να μην καταστραφούν για να προωθηθεί το εμπόριο. Ε, θα χρειαστούν λοιπόν επαρκείς πόροι κατά τρόπον ώστε συμφωνία να μπορέσει να εφαρμοστεί ικανοποιητικά. Σχετικά με την Λιβερία έχουμε χαιρετήσει όπως θα θυμούνται οι συνάδελφοι ε, την κίνηση της Λιβερίας κατόπιν ε, του εμφυλίου πολέμου της δεκαετίας του 90 όπου ένα μεγάλο μέρος του τροπικού δάσου υπήρχε ε, ξεθύματο των ε, διαμαχών και είναι πολύ θετικό ότι τώρα η χώρα έχει λάβει αυτή την ε, θέση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να παρακολουθούμε ε, τις εξελίξεις και στις δύο χώρες αυτές και να προσέξουμε πώς θα εφαρμοστεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την ξυλία το 2013 κατά κατά τρόπον ώστε να υπάρξει σωστή παρακολούθηση. Ναι, υπάρχουν και παρεμφερείς ε, συμφωνίες οι οποίες όπως είπατε έχουν ήδη ισχύσει για την Κάνα, το Κονγκό και το Καμερούν. Ο επόμενος ομιλητής, επίσης σκιώδης εισηγητής, είναι η Κάθριν Πιέρντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την προσπάθεια αυτή ρύθμισης και προστασίας των φυσικών περιοχών του κόσμου τις οποίες φαίνεται ότι παίζουν πάρα πολύ. Πέρσι ήμουν στο Καμερούν και επισκέφθηκα μία περιοχή ξυλία στην οποία παράνομα φόρτωνε ξυλία στρατό. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν όλε αυτέ οι συμφωνίε και να έρθουν σε ισχύ για να εξασφαλίσουμε ότι πραγματικά οι χώρε αυτέ την χάνουν των κατάλληλων συμφωνιών για αυτά τα, για αυτά τα οποία παρέχουν. Θα πρέπει όμως να τεθούν σε εφαρμογή και όχι να παραμείνουν μόνο επί χάρτου. Όσον αφορά την ε, συμφωνία με την Ενδονησία άκουσα σε διάφορες εκθέσεις ότι μεταφέρουν τροπική ξυλία σε πολύ μεγάλες ποσότητες προς την Ιαπωνία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με τους Ιάπωνες για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και είναι ότι κάνουν εντελώς αντίθετο προς τις συμφωνίες. Κάτι άλλο το οποίο με απασχολεί είναι η έκθεση για ε, τα διάφορα ε, υποπροϊόντα ξυλίας, δηλαδή ε, τα κομματάκια ξυλού τα οποία χρησιμοποιούνται, τα wood chips, τα οποία χρησιμοποιούνται ε, ως καύσιμο στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε όλα αυτά τα υποπροϊόντα ξύλου, από τι είδους ξυλία προέρχονται. Με απασχολεί αυτό. Ευχαριστώ. Από τους πράσινους ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές παρατηρήσεις έγιναν από τον Ντέιβιτ. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε επιβάλει το εμπάργκο για την εξαγωγή ξυλίας από την Λιβερία. Η εξελίξη στη Λιβερία είναι ενδιαφέρουσες. Πρόκειται για μία από τα... Πρόκειται για περιοχή η οποία έχει ένα από τα πιο σημαντικά βάσεις στην περιοχή της Αφρικής. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω κάτι που ανέφερε ο Ντέβιτ και για τους αυτόχθονες στα πλαίσια της ε, περιοχής αυτής της λεκάνης στο Κονγκό και το τι γίνεται με την ξυλία. Η πρώτη παρατήρηση προς τη γητήρια είναι η εξής. Τελευταία φορά για το Καμερούν και το Κονγκό κατορθώσαμε να κάνουμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια και νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό να μπορέσουμε να το συζητήσουμε παρουσία της Επιτροπής του Συμβουλίου στην Ολομέλεια ώστε να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να, να νομιμοποιήσουμε και να κάνουμε πιο επίσημε τις αποφάσεις που θα πάρουμε στο τέλος της συζήτησής μας. Όσον αφορά τώρα την Κομισιόν. Μετά από την έγκριση συμφωνία του Καμερούν και το Κονγκό υπήρχε μια δέσμευση εκ μέρου τη Επιτροπής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις συμφωνίες Φλέκ και κυρίως για την ε, συμμετοχή του συνόλου των φορέων εκ μέρους της, πολι... της κοινωνίας των πολιών, πολιτών και να τους δώσει την δυνατότητα να κάνουν κάποιες κρίσεις και επικρίσεις όταν υπάρχουν προβλήματα είχε εκφράσει αυτή τη βούληση η Κομισιό. Κατά κάποιο τρόπο πλατείασε η όλη διαδικασία. Θα ήθελα να μας πει η Κομισιό. Είναι διατεθειμένη να αναλάβει την δέσμευση να ε, συμμετέχει εκ του σύνεγγυς περισσότερο στα τέτοιου είδους θέματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Τελικά ο Χέλμουτ Σόλτς από την Γουε Ευχαριστώ Πρόεδρε. αντικαθιστώ τον σκιάδη συγητή μας που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Μου ζήτησε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχέση με την έκθεση αυτή. Υποστηρίζει τη γενική θέση της κυρίας Κάσκεμ ο συνάδελφος και χαιρετίζει την προσέγγιση της. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε βήμα μπορεί να ληφθεί για να καταπολεμήσουμε την ε, ε, αποψήλωση των δασών στην περιοχή και την παράνομη υλοτομία. Επίσης, ο συνάδελφος εκφράζει ανησυχίες για το τι ακριβώς γίνεται στην Λιβερική. Μας υπενθυμίζει ότι η Λιβερία είχε πρόβλημα ε, εθνικό, εσωτερικό πριν από το 2003 και υπήρχε πρόβλημα με την εκμετάλλευση ε, διαφόρων πόρων της και κυρίως ξηρίας. Τώρα, ξέρουμε ότι η εκ του παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων, τοπικό επίπεδο, και όλων όσων συμμετέχουν στη συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να ζητήσει από την Επιτροπή αν επαρκεί. Να ζητήσουμε από την Επιτροπή να παρακολουθεί την ε, κατάσταση για να μας κάνει έκθεση και αν δεν θα πρέπει να ζητήσουμε εμείς από το Κοινοβούλιο μια ετήσια έκθεση για τις εξελίξεις. Επίσης, το 85% του πληθυσμού της Λιβερίας βρίσκεται κάτω από το κατόφλι της φτώχειας, ιδιαίτερος τα άτομα αυτά πολλές φορές χρειάζεται για να μπορέσει να επιβιώσει η οικογένεια να καταφύγουν σε τέτοιου είδους ε, παράνομες δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι γίνεται σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης χώρας και κυρίως τι γίνεται όπως υπενθύμησαν και οι άλλοι σχεδόν και ο Ντέβιτ Μάρκεν με τον ε, πληθυσμό της Λιβερίας για να ξέρουμε αν θα γίνει αλλά εν πάση θα κατατεθούν και οι σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε η κυρία Φάλκονερ από την Επιτροπή ο κύριος Μπλίνεβα ποιος είναι εδώ, συλλάβει το λόγο.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 Ευχαριστώ. Ο Ζων Μπρινδάν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για το ενδιαφέρον της για αυτές τις συμφωνίες και τη στήριξη για αυτές τις δύο συμφωνίες. Σημειώνουμε τη σύσταση της Επιτροπής και ε, τα συμπεράσματα της επεξηγηματικής, ε, του επεξηγηματικού σημειώματος σχετικά με την Κεντρική Αφρική ε, για του ε, τοπικό πληθυσμό που αναφέρθηκε στη διαπραγμάτευση. Η ε, πληροφορία που μπορώ να σας δώσω σήμερα είναι ότι καταρχήν η κυβέρνηση της Κεντρικής Αφρικής μελετά και μάλιστα και ε, ε, σκοπεύει να υπάρξει ανάθεση ε, κοινοτικών δασών και να υπάρχουν κείμενα τα οποία θα αναφέρουν άμεσα τα συμφέροντα του τοπικού πληθυσμού. Όσον αφορά την χρηματοοικονομική ενίσχυση, όντως χρειάζεται να υπάρξει εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ενώσης ενώ η συμφωνία δεν προβλέπει δέσμευση οικονομική στήριξης και πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει 6,7 εκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή του προγράμματος πέραν της στηρίξεως των προγραμμάτων της τοπικής κοινωνίας και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα αλλά χρειάζεται στήριξη των κρατών μελών για να μπορέσει να υπάρξει μία πλήρης εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Δηλαδή είναι απαραίτητη η στήριξη των κρατών μελών για να εφαρμοστούν τα ΦΛΕΚΤ όσον αφορά τη θεματολογία της αποψηλώσεως των δασών και της αύξησης του διοξιδίου του άνθρακο σε σχέση με την αποψήλωση των δασών και την εφαρμογή των φλέκτ εξετάζουμε το πρόβλημα προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί κανείς να πατάξει αυτή την καταστροφή των δασών όταν δεν υπάρχει ε, σωστή δασική διαχείριση η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με ε, την καταπολέμηση των ε, κλιματολογικών αλλαγών και δίνω το λόγο τώρα στη συνάδελφό μου Τζούλια Φάλκονερ για περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Συμμετείχα στις συζητήσεις με την Λιβερία για τα τελευταία 7 χρόνια. Νομίζω ότι ε, τα σημεία που επισημάνθηκαν για τη συμφωνία με τη Λιβερία ήταν ε, πολύ σκόπιμα. Υπάρχει ένα επίπεδο δέσμευσης ε, από την ηγεσία της λιβερικής κυβέρνησης, εν μέρη λόγω της ιστορίας της, λόγω του επιβαρημένου ιστορικού της Λιβερίας με τον εμφύλιο πόλεμο. Ο συγκεκριμένο ε, τομέα είναι πολύ σημαντικός ε, στη Λιβερία και ως τμήμα της διαδικασίας ανοικοδόμησης της Λιβερίας. Τώρα, για τον τρόπο που προσέγγισε η κυβέρνηση αυτέ τις διαπραγματεύσεις ε, και τη διαβούλευση με άλλα ενδιαφέροντα μέρη ήταν πραγματικά παραδειγματικό. Οι πραγματικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή στη Λιβερία βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά την ικανότητα και προσπαθούμε να προγραμματίσουμε την στήριξή μας για να τους παράσχουμε τους απαραίτητους πόρους. Έχουμε προς το παρόν πρόταση για 10 εκατομμύρια από την Επιτροπή, περαιτέρω πόρους από τον Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα κράτη-μέλη. Και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε ε, τη διαδικασία και να μπούμε στη φάση εφαρμογής πολύ σύντομα. Η πρώτη κοινή συνεδρίαση μετά την εφαρμογή θα λάβει χώρα στα τέλη Μαρτίου στη Λιβερία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε όμως ότι ε, παίρνει πολύ καιρό να περάσουμε από την υπογραφή της σύμβασης στην ε, πρακτική της εφαρμογή. Πρέπει να ολοκληρωθεί η δικασία κύρωσης και στις δύο πλευρές. Τα όσα αναφέρθηκαν για την ενημέρωση του Κοινοβουλίου τα σημειώνουμε. Η κάθε συμφωνία συνοδεύεται και από ε, δέσμευση ενημέρωσης, σίγουρα σε ό,τι αφορά την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες δημοσιεύονται, και ενημέρωση για όλες τις ε, κοινέ ε, αποστολές παρακολούθησης. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή αν θέλετε να ζητήσετε επικαιροποιημένες πληροφορίες. Ίσως ε, στο πλαίσιο και τη συζήτηση στην Ολομέλεια, αν αυτό κανονιστεί. Όμως πρόθεσή μας είναι να σας ενημερώνουμε. Ευχαριστώ. Ακόμα έχουμε χρόνο για... Ε, συγγνώμη, μάλλον παίρνουμε χρόνο από την ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Επομένω, ε, ο εισηγητή έχει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλου του συναδέλφου για τα σχόλια και για τις απόψεις που διατύπωσαν. Είμαι διαθέσιμη ε, να συνεχίσω να συζητώ τα διάφορα θέματα και πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό το ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει υπέρ του πληθυσμού διότι η Λιβερία μέχρι το 2003 ε, ήταν σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου και αν δούμε πόσο θετικές εξελίσεις έχουμε τα τελευταία χρόνια ε, ε, είναι εκπληκτικό διότι εμείς χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο για να εφαρμόσουμε διαδικασίες και πιστεύω ότι εδώ είμαστε στο σωστό δρόμο και όσον αφορά τους άλλους σκιώδεις εισηγητές πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει στην Ολομέλεια συζήτηση και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι ε, ενδιαφέρθηκαν και ε, μας ε, διέθεσαν τον χρόνο που χρειαζόμασταν. Ευχαριστώ. Η ε, προθεσμία για τροπολογίες είναι μέχρι τις 6 Μαρτίου 6 το απόγευμα και η ψηφοφορία όπως έχει προβλεφθεί θα διεξαχθεί στη συνεδρίαση τέλος Μαρτίου διότι δεν υπάρχει ακόμη διότι δεν υπήρχε μεν ακόμη αλλά έχει τώρα κατατεθεί το έγγραφο που μας έλειπε από το Συμβούλιο προς το Κοινοβούλιο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και χωρίς χρονοτριβή προχωρούμε ε, εις ε, την ε,